κύριε Πρόεδρε και σας δίνω απευθείας το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας, ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Προπύργιου της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να μοιραστώ μαζί σας το όραμα μας για την Ένωση και για να παρουσιάσω τις κύριες προτεραιότητες της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. Εκφράζω τον βαθύ σεβασμό και τα συγχαρητήρια μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο που διαδραματίζει στην υπεράσπιση και την προοή των θεμελιωδών αρχών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτρέψτε μου δε να υπογραμμίσω την δική μου προσωπική ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει καταστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθέτη μαζί με το Συμβούλιο για τους πλήστους νομοθετικούς φακέλους. Αναμφίβολα η θετική αυτή εξέλιξη ενισχύει και διευρύνει τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, η Κύπρος αναλαμβάνει για πρώτη φορά την εξαμηνία Προεδρία του Συμβουλίου από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την Ένωσή μας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση ταλανίζει κρατημέλη, ενώ τη μεγαλύτερη πίεση εξακολουθεί να δέχεται η Ευρωζώνη. Αναντίλεκτα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση μας απαιτούν ρηξικέλευθες ευρωπαϊκές απαντήσεις. Έφτασε ίσως η ώρα να στραφούμε για καθοδήγηση στην αφεντηρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, τότε που μέσα από τις τάχτες του πολέμου τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Είναι η ώρα που θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και θάρρος και την προνοητικότητα από το θάρρος και την προνοητικότητα των πατέρων του ευρωπαϊκού οράματος. Ενός οράματος ειρήνης, δημοκρατίας, πλουραλισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε τέτοιες περίοδους κρίσεων καθίσταται πιο επιτακτική η ανάγκη για να πετύχουμε μια πιο αλληλέγγυα και αποτελεσματική ένωση, μια καλύτερη Ευρώπη. Το χρωστάμε στους οραματιστές της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μα κυρίως το χρωστάμε στους νέους μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η επίτευξη μιας καλύτερης Ευρώπης αποτελεί καθολικό αίτημα των πολιτών της Ένωσης. Εμείς έχουμε υποχρέωση να αφουγκραστούμε τους πολίτες μας και να καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων μας για μια Ένωση που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της. Μια Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής της ευημερίας, της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Ακούραστα θα εργαστούμε κατά το τρέχον εξάμεινο για να προωθήσουμε ακριβώς εντός του Συμβουλίου και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που θα συνδράμει στο στόχο μιας κοινωνικά αλληλέγγυας και αποτελεσματικής Ευρώπης. Μιας Ένωσης με πιο όρατα ωφέλη για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι ο γενικότερο πολιτικός μας στόχος κατά το εξάμεινο της Κυπριακής Προεδρίας και πραγματικά ευελπιστούμε όπως έχουμε στην προσπάθεια μας αυτή την στήριξη και την αρρωγή όλων των θεσμικών οργάνων και ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει περάσει μέσα από πολλές κρίσεις από τη σύστασή του. Φαίνεται όμως πως η συνεχιζόμενη κοινωνικο-οικονομική κρίση, απότοκο σε μεγάλο βαθμό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αποτελεί την μεγαλύτερη συγκριτικά πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει από την ίδρυση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί έχει απειληθεί σημαντικά η ευημερία και η κοινωνική συνοχή στην Ένωση. Παράλληλα έχουν παρατηρηθεί ρήγματα στην θεσμική ενότητα της Ένωσης λόγω και των διαφορετικών προσεγγίσεων που ακολουθήθηκαν ως προς τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν με άμεση προτεραιότητα την σταθεροποίηση της κατάστασης. Πιστεύω ακράδαντα πως αποτελεί ανάγκη η στήριξη της συνοχής και της ενότητας των κρατών μελών. Μαζί μπορούμε σίγουρα να τα καταφέρουμε καλύτερα. Είμαι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεπεράσει με επιτυχία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εξέλθει χειρότερη τη τρέχουσα κρίση. Μια κρίση που δυστυχώ κλονίζει σε μεγάλο βαθμό και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο θεσμικό οικοδόμημα μας. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όμω με επιτυχία τι προκλήσεις εάν επιδείξουμε συλλογικά την απαραίτητη εμπιστοσύνη στους κοινού ευρωπαϊκούς θεσμούς στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η κοινοτική μέθοδος έχει αποδειχτεί διαχρονικά ισχυρό όπλο στην προάσπιση των κοινών μας συμφερόντων και θα πρέπει με κάθε τρόπο να προστατευτεί. Η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης που να στηρίζει την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή αποτελεί κατά την άποψή μου την καλύτερη οδό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρέχουσας κοινωνικο οικονομικής κρίσης. Αγαπητοί φίλοι, θεωρώ ότι για να έχουμε Θεωρώ ότι για να έχουμε επιτυχή θεραπεία των πληγών που, έχουν προκαλέσει, που έχει προκαλέσει η κρίση, θα πρέπει ταυτόχρονα να προβούμε και στη σωστή διάγνωση για τα αίτια που τις προκαλούν. Θα πρέπει από κοινού να κάνουμε μια τολμηρή και σε βάθος ανάλυση της ουσίας και του εύρους της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να προβούμε ακόμα και σε αυτοκριτική, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την πιθανή πολιτική αδράνεια ή τις αδυναμίες των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη τις περασμένες δύο δεκαετίες. Κυρίως τις περασμένες δύο δεκαετίες. Δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός πως οι πολιτικές που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια προβάλλοντας ένα μοντέλο απόλυτης και δογματικής αγκίστρωσης στην ελευθερία της αγοράς χωρίς κανένα κοινωνικό και κρατικό έλεγχο έχουν αποτύχει. Γιατί πολύ απλά ένα πράγμα είναι η ελεύθερη κοινωνική οικονομία της αγοράς και άλλο βεβαίως η ασυδοσία των αγορών, ελλείψη κρατικής εποπτείας, και συναφών ασφαλιστικών δικλείδων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να καταστούν οι κοινωνίες μας έρμεο των αγορών και των ιδιωτελών συμφερόντων που τις χειραγωγούν. Αποδείχτηκε δε εκ των πραγμάτων πως τα όποια μέτρα λήφθηκαν τα περασμένα χρόνια υπήρξαν αναποτελεσματικά ένεκα της ανάλυσης της κρίσης με βάση την πεπατημένη που μας θέλει να ενοχοποιούμε μόνο τους κερδοσκόπους και κάποτε τις αγορές. Οι πολιτικές αυστηρής λιτότητας που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης όχι απλά αποδεικνύονται ανίκανες να επιλύσουν τα προβλήματα, αλλά τα επιτείνουν. Με τις πολιτικές λιτότητας και μόνον ξυλώνεται το κοινωνικό κράτος και καθυλώνεται η ανάπτυξη. Η οικονομία και η αφόρος ανάπτυξη πρέπει να εξυπηρετούν την κοινωνία – ο παραγόμενος πλούτος πρέπει να καταμερίζεται πιο δίκαια. Δεν μπορεί η προσέγγιση να είναι κοινωνικοποίηση των ζημιών και ιδιωτικοποίηση των κερδών. Δεν γίνεται να φορτώνουμε με τις πολιτικές μας το βάρος της τρέχουσας κρίσης στους ώμους όλων εκείνων που με τα βίας βγάζουν τα προστοζήν. Οι απλοί πολίτες των κρατών μελών της Ένωσης είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται για τις εγγενείς αδυναμίες που όπως αποδείχτηκε βαρύνουν τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ηθική και πολιτική υποχρέωση να καταμεριστούν δίκαια τα βάρη από την κρίση και σίγουρα θα πρέπει να προστατευτούν τα οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού. Επιτρέψτε μου αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, να εκφράσω στο σημείο αυτό τον βαθύ συγκλονισμό που αισθάνομαι κάθε φορά που στους δέχτες των τηλεοράσεων μας βλέπουμε εικόνες δυστυχίας, με ουρές πολιτών να συνοστίζονται σε κοινωνικά συσσίδια για να εξασφαλίσουν μια μερίδα φαγητού, ουσιαστικά μια μερίδα επιβίωσης είναι το λιγότερο προσβλητικό για όλους μας να ανεχόμαστε μια τέτοια κατάσταση στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να μένουμε ατάραχοι βλέποντας την φτώχεια να οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και εξαθλίωση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Ευρώπης. Από αυτό το επίσημο βήμα σας καλώ φίλε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εργαστούμε από κοινού για να εξεύρουμε τρόπους διεύρυνση και παράλληλη ενίσχυση του προγράμματο επιστημιστικής βοήθεια για του άπορους συμπολίτε μας χρησιμοποιώντας γεωργικά προϊόντα παρέμβαση. Θα είμαι πραγματικά ο ευτυχέστερο των Ευρωπαίων αν μέχρι το τέλο τη Κυπριακή Προεδρίας καταφέρουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα επί του εν λόγω προγράμματο, υιοθετώντα ή υιοθετώντα άλλε παραπλήσιες δράσεις ισόποσου αποτελέσματο στη βάση των νομοθετικών πρωτοβουλειών της Επιτροπής, περιορίζοντας έτσι όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως δεν επιλύεται με αυτόν τον τρόπο. Το μείζον επομένως, κατά τη δική μου άποψη, αποτελεί η δικαιότερη ανακατανομή του παραγόμενου εισοδήματος. Μια συνεπής και πιο ανθρωποκεντρική κοινωνική πολιτική που σε συνδυασμό με την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Τη ραχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκή οικονομία θα οδηγήσει σε περισσότερη απασχόληση και στην πολυσυζητημένη κοινωνική συνοχή εντό της Ένωσή μα. Αναντίλεκτα, ιδιαίτερα το τελευταίο έτος, με τη συμβολή όλων και κυρίω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν προωθηθεί δράσει που θα επιταχύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη για την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δράσεις που αναμένουμε ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης πρωτίστως των νέων και σε μια πιο πράσινη οικονομία. <clears throat> και όλα αυτά συμπληρωματικά των μέτρων που λήφθηκαν κατά προτεραιότητα προς αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να υπάρξει μια συμφιλίωση αφενός της προσέγγισης για δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί ναι είναι σημαντικό να περιορίσουμε τις σπατάλες και να νοικοκυρέψουμε τα δημόσια οικονομικά και αφετέρου της προσέγγισης για υλοποίηση μιας ισχυρής στρατηγικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Ως Προεδρία του Συμβουλίου Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία μαζί σας, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσουμε δράσεις που θα στοχεύουν στην μίκρυνση της κοινωνικής πίεσης που έχει δημιουργηθεί σε πλήστες τόσες χώρες της Ένωσης μας και που δυστυχώς πλήττει τις περισσότερες φορές τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, το μέλλον της Ευρώπης μας. Περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, αυτό χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Μόνο έτσι θα κάνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να πιστέψουν ξανά στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Μόνο έτσι θα μειώσουμε το χάσμα που χωρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες από τα απρόσωπα και απόμακρα πολλές φορές για αυτούς κέντρα λήψης των αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, μέσα ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο της προσπάθειας για μια καλύτερη Ευρώπη, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτη προτεραιότητα, μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική και βιώσιμη. Η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 με απότερο σκοπό την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποδοτικού προϋπολογισμού της Ένωσης που να οδηγεί στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Η Προεδρία θα προσπαθήσει να πετύχει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις κοινέ πολιτικές της προγραμματικής περίοδου όπως η κοινή γεωργική και αλλιευτική πολιτική, η πολιτική συνοχής, και οι πολιτικές της έρευνας και καινοτομίας. Ιδιαίτερη σημασία είναι η ενεργειακή πολιτική, καθώς και η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, τα οποία θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και στην περαιτέρω ολοκλήρωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελέσει σημαντικό θέμα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με γνώμονα την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στις πολιτικές των μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επανενεργοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης. Θα γίνει ειδική διάσκεψη στη Λεμεσόν με την παρουσία και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αποφασιστεί, θα εγκριθεί ειδική διακήρυξη για το θέμα. Δεύτερη προτεραιότητα, μια Ευρώπη με πιο αποδοτική οικονομία βασισμένη στην ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερη αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ένωσης η προεδρία θα αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής ευρώπη. 2020. επιπρόσθετα η ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης και η προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης είναι μείζονος σημασίας για την κυπριακή προεδρία. οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτελούν επίσης σημαντικό θέμα στο πρόγραμμα μας καθώς θα συνεισφέρουν στην προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και με την ευκαιρία της 25 ης επαιτίου της ενιαίας αγοράς θα, επίσης, θα προωθηθεί επίσης η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς με στόχο να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και στήριξη στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Αναμφίβολα η ενιαία αγορά αποτελεί τη σταθερή βάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδιαίτερα εν καιρό οικονομικής κρίσης χρειάζεται να βελτιώσουμε την ενιαία αγορά δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Τρίτη προτεραιότητα, μια Ευρώπη που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή. Μια από τις σημαντικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους στόχους για την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόθεσή μας είναι να αξιολογήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιδιώξουμε να χαρτογραφήσουμε την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην διεργασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η κοινωνική συνοχή αποτελεί σημαντική πτυχή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ουσιώδη στόχο των προσπαθειών για την αποτελεσματική έξοδο από την κρίση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας της Κυπριακής Προεδρίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής θα επικεντρωθούμε στη συνέχιση της εργασίας για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και ειδικότερα την πρόθεση της ευζοίας των παιδιών. Με την ευκαιρία δε του έτους ενεργούς γύρανσης η Κυπριακή Προεδρία θέλει να προβάλλει το μήνυμα πως η ενεργός γύρανση δεν περιορίζεται μόνο στην απασχόληση, αλλά περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων σε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτιακά δρόμενα. Σε ό,τι αφορά στα θέματα της ισότητας, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει την εργασία για την διαμόρφωση δικτών για την βία ενάντια στις γυναίκες και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε υπηρεσίες στήριξης θυμάτων. Η Προεδρία θα εμβαθύνει επίσης συζητήσεις, θα ενθαρρύνει με συγχωρείτε, επίσης συζητήσεις σχετικά με το πρόβλημα του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Ένας από τους κύριους στόχους της Προεδρίας θα είναι επίσης η δημιουργία του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012 με την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών για την προστασία των δικαιωμάτων όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν οι διαπραγματεύσεις για τα προγράμματα της επόμενης γενιάς εράσμους φορόλ και προώθηση του αλφαβητισμού. Τέταρτη προτεραιότητα, η Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονες της. Η Κυπριακή Προεδρία θα έχει στενή συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Στο πλαίσιο αυτό και εν ώψη των σημαντικών πολιτικών ανακατατάξεων που λαμβάνουν χώρα στην νότια ακτή της Μεσογείου, ιδιαίτερη βαρύτητα θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί στη νότια διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, προωθώντας τις σχέσεις της Ένωσης με τις μεσογειακές χώρες. Για μένα τουλάχιστον είναι αυτονόητο πως οι αραβικοί λαοί της νότιας γειτονίας μας που ξεσηκώθηκαν και επιζητούν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα πρέπει οι ίδιοι να επιλέξουν μέσα από μια ελεύθερη και συμμετοχική διαδικασία το καθεστώς διακυβέρνησης τους. Αποτελεί στρατηγικό λάθος, κατά τη γνώμη μου, να επιχειρήσει η Ευρώπη να επιβάλλει σε αυτούς τους λαούς το δικό της μοντέλο δημοκρατίας. Αυτό όμως που η Ευρώπη μπορεί και οφείλει να κάνει είναι η στήριξη του οράματος των νέων που εκφράζουν το αραβικό όραμα για δημιουργία πλουραλιστικών κοινωνιών, θεμελιώδες στοιχείο των οποίων να αποτελεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει τα απαιτούμενε διεργασίε σχετικά με την διαδικασία διεύρυνσης και που πράγματι αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ένωσης. Φίλε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση μου κάνοντας μια πολύ σύντομη αναφορά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία που ομολογουμένως αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα επί του οποίου εδράζεται η κοινή μας ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Στην πολιτεία του πλάδωνα ο μεγάλος φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο Σοκράτης, ρωτάται ποιο είναι το νόημα της ζωής και ο Σοκράτης απαντά ευθέω το να είσαι καλός Αθηναίος. Και τι είναι Σοκράτη ο καλός Αθηναίος, ρωτάει ξανά ο Πλάτωνας. Η απάντηση αγαπητοί φίλοι ήταν απλή αλλά γεμάτη διαχρονικό νόημα και σκοπό. Ο καλός Αθηναίος είναι αυτός που αφήνει την Αθήνα καλύτερο μέρος από ό,τι τη βρήκε. Πολύ απλά, πολύ σωστά και πολύ ωραία. Η Αθήνα του Σοκράτη και του Πλάτωνα είναι βεβαίως σήμερα το κοινό απόκτημα μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ηγέτες της Ευρώπης έχουμε καθήκον να εργαστούμε ακούραστα για να κάνουμε την Ευρώπη μας ένα καλύτερο μέρος για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως για τις μελλοντικές γενναίες με καινοτόμε και ρηξικέλευτε πολιτικέ που θα έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τι εύλογε του ανάγκε, μπορούμε να επιτύχουμε αηφόρο οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Όπω ακούσατε και από τι προτεραιότητε που μόλι ανέφερα, η Κυπριακή Προεδρία έχει καταρτήσει ένα ομολογουμένω φιλόδοξο πρόγραμμα. Έχουμε πάντω επίγνωση τη ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία καθώς και των προκλήσεων που τίθενται ενώπιον μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως βέβαια γνωρίζετε, η χώρα μου αντιμετωπίζει μια επιπρόσθετη πρόκληση λόγω του προβλήματος της αναχρονιστικής διέρεσης εξαιτίας της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής του βόρειου τμήματος του νησιού. Θα ήθελα όμως κατηγορηματικά να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφησούμε προσπαθειών και δεν θα επιτρέψουμε στα προβλήματα που τυχόν αποπειραθεί να δημιουργήσει η κατοχική δύναμη να μας αποπροσανατολίσουν από την ενάσκηση μιας καθόλου ευρωπαϊκής προεδρίας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κυπριακή Προεδρία θα προσπαθήσει να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεων και των αρμοδιοτήτων της στην επίτευξη μιας καλύτερης Ευρώπης προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Στους έξι μήνες που έχουμε μπροστά μας, μπορούμε με τη βοήθεια και τη στήριξη όλων σας, θεσμικών παραγόντων, της κοινωνίας των πολιτών και βεβαίως εσάς, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συμβάλλουμε σημαντικά στην επίτευξη αυτού του μεγάλου κοινού μας στόχου. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Χριστόφια. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πρόεδρο Ζωζέ Μανέλ Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε τη Κυπριακή Δημοκρατία, αξιότιμα μέλη. Καταρχά, να εκφράσω προ τον Πρόεδρο Χριστόφια και την Κυπριακή Προεδρία τη δική μου και την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πλήρη υποστήριξη για την Προεδρία του Συμβουλίου. Θα συνεργαστούμε στο πνεύμα πλήρους συλλογικότητας σας ευχόμαστε κάθε δυνατή επιτυχία προς το συμφέρον της χώρας σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Η Προεδρία του Συμβουλίου είναι προφανώς μια πρόκληση και για μεγάλες και για μικρές και για παλαιότερα και για νεότερα κράτη-μέλη. Και φυσικά οι προκλήσεις αυτές διπλασιάζονται όταν ασκείται την Προεδρία για πρώτη φορά στην σημερινή οικονομική συγκυρία του, του λεχθέντος έχω κάθε εμπιστοσύνη στην ε, ετοιμότητα να αναλάβει η Κύπρος αυτήν την μεγάλη ευθύνη. Και βεβαίως ε, το επιβεβαίωσε αυτό η ομιλία του Προέδρου Χριστόφια, η δέσμευσή του για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή μέθοδο. Οι προπαρασκευές τους άρχισαν εδώ και τρία χρόνια σχεδόν. Ε, εν τω μεταξύ, οι Κυπριακές ε, Αρχές και η Επιτροπή σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο συνεργάστηκαν καρποφόρα μαζί αύριο και μεθαύριο. Οι κοσμήτορες θα συναντηθούν με την ομάδα της Προεδρίας στη Λευκοσία όπου θα εκφράσω την εκτίμησή μας για τον ιδιαίτερα ικανό τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκαν. Μετά λοιπόν την έναρξη πρέπει να συνεχίσουμε φυσικά την εργασία μας, την έναρξη της Προεδρίας και εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι σωστά αντιλαμβάνεται η Κυπριακή Προεδρία τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπίσει. Συμμεριζόμεθα τους στόχους της Προεδρίας για μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη που να βασίζεται σε βιώσιμη ανάπτυξη, αλληλεγγύη, χωρίς αποκλεισμού, που να παίζει μεγάλο ρόλο στο παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην ε, γειτονία της. Οι στόχοι αυτοί απαιτούν δράσεις που να εντάσσονται στην ε, τριμερή λογική που εδώ και πολύ χρόνο υποστηρίζει η Επιτροπή και που πρέπει να είναι η βάση της εργασίας μας. Πρώτα απ' όλα η οικονομικά, βαθιέ ε, διαρθρωτικέ αλλαγέ και στόχο προσιλωμένε επενδύσει. Με βάση αυτού του τομεί και μεγιστοποιώντα την επίπτωσή του, θα έχουμε μια επιτυχή Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου. Για να είναι επιτυχή σε Προεδρία, πολύ σημαντικό θα είναι να στοχεύσουμε τι ε, νομοθετικέ πρωτοβουλίε κλειδιά, όπου μπορούμε να πετύχουμε απτή πρόοδο μέχρι τέλο του χρόνου. Πρώτο και κύριο έχουμε το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα από τα κύρια όργανά μα για να υπάρξουν επενδύσεις που να προσθέτουν αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για να υπάρξει ανάπτυξη και θέση εργασία στην Ευρώπη. Ο πρόεδρο Χριστόφια, ο πρόεδρος Σούλτ, κύριε πρόεδρε Χριστόφια, κύριε Σούλτ, αξιότιμα μέλη, να σκάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει συμφωνία για το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι τέλο του χρόνου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά είναι εφικτό. Αυτό θα αποστείλει σαφέ μήνυμα ότι όταν πρόκειται για θέματα ανάπτυξη, θα αναλάβουμε δράση όχι μόνο λόγια. Εάν επιτύχουμε αυτό το στόχο μέχρι τέλο του χρόνου, όχι οποιοδήποτε συμφωνία, αλλά μια καλή, μια πολύ καλή συμφωνία, θα σημάνει ότι θα παράσουμε μια μεγάλη υπηρεσία σε όλου του πολίτε τη Ευρώπη. Θα είναι μια επιτυχία και για την Κυπριακή Προεδρία. Η Επιτροπή τις επόμενε μέρε θα υποβάλει ενημερωμένα ε, χρηματοοικονομικά στοιχεία για την πρότασή μα για το πολιτέ δημοσιονομικό ε, πλαίσιο που θα συμπεριλάβει και την επίπτωση της ένταξης της Κροατίας το 2013 λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία εθνικά και περιφερειακά στατιστικά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές θα είναι αρκετά περιθωριακές στο συνολικό ποσό, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η ενημέρωση για να υπάρχει ακρίβεια, διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση. Οπότε η Προεδρία με αυτή τη βάση θα μπορέσει να προπαρασκευάσει τις σοβαρές συζητήσεις και για συγκεκριμένα νούμερα από το φθινόπωρο. Επαναλαμβάνω αυτό που ήδη είπα τα στοιχεία που προτείναμε πέρσι εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως. Είναι τα σωστά, είναι ρεαλιστικά στοιχεία. Και είναι ε, μια απόδειξη ρεαλισμού, αλλά και αρκετή φιλοδοξίας στη σημερινή συγκυρία. Καλό λοιπόν και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν ότι αυτά που προτείναμε ήδη είναι μια πολύ καλή βάση για ένα συμβασμό. Φυσικά ε, οι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πακέτο μαζί με το συνολικό πλαίσιο. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να καταλήξουν και για τις κλαδικές προτάσεις για τους κυρίους τομείς πολιτικής, που είναι η βάση της προσπάθειάς μας για να υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Παράλληλα λοιπόν, πρέπει να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος για την νέα γενιά των διαφορετικών ταμείων, τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑΓΑΜΑΠΗ, την κοινή αλληλευτική πολιτική, τον ορίζοντα 2020 για την έρευνα και την ε, καινοτομία, την δυνατότητα συνδυασμού της ε, σύνδεσης της Ευρώπης και τα διευρωπαϊκά δίκτυα και επίσης και τα εξωτερικά οικονομικά μας μέσα είναι σημαντικά. Συνολικά λοιπόν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και περίπου 70 κλαδικά προγράμματα, τομεακά προγράμματα είναι μεγάλη πρόκληση να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Μεγάλη προσπάθεια από πλευρά Προεδρία του Συμβουλίου. Μια προσπάθεια που εμεί ω Επιτροπή θα υποστηρίξουμε πλήρω. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι μόνο ένα από του μοχλού για ανάπτυξη και θέσει απασχόληση. Υπάρχουν και άλλες κρίσιμες ε, πολιτικέ όπου πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Καλωσορίζω ότι ο πρόεδρος Χριστόφια συμφωνεί μαζί μου ότι πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο όλα τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Κοινοβουλίου, του επόμενου μήνε. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να επιτύχουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, αποτελέσματα που να είναι σταθερά, δεσμευτικά και να μην εξαρτώνται από τις εξελίξεις μετά τη λήψη τους. Θα συνεχίσουμε την εργασία μας για την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν και περισσότερες ενέργειες για την προώθηση με ταχεία διαδικασία νέων νομοθετημάτων για την ε, ενιαία αγορά. Αυτό που λέμε η πράξη ενιαία αγορά. Έχουμε ήδη την πράξη ενιαία αγορά 1. Θέλουμε τώρα να περάσουμε την πράξη ενιαία αγορά 2. Ελπίζω η Προεδρία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση και σε ευχαριστώ πολύ για την ισχυρή δεσμευσή σας για την ανάγκη να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά, Πρόεδρε Χριστόφια. Πρόεδρε Αξιότιμα Μέλη, όπως είπα και χθε ενώπιον σας, θα συνεχίσουμε έντονες προσπάθειες για τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό χώρο και θα υποβάλουμε γι' αυτό νέες προτάσεις που αφορούν τα πρώτα βήματα για να δημιουργήσουμε αυτό που αποκαλούμε μια τραπεζική ένωση. Δηλαδή να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για τις τράπεζες ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με βάση το άρθρο 127 της συνθήκης. Και την ίδια στιγμή θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την συνολική αρχιτεκτονική της ε, ε, Ευρώπης 27, σύντομα 28, ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική της ενιαίας αγοράς, ούτως ώστε να εγγυηθούμε την ακαιρεότητα της Ένωσής μας και φυσικά πλήρη δικαιώματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τις ηθίκες. Πολλά πρέπει να κάνουμε για να οικοδομήσουμε με βάση τις ε, ε, προτάσεις που έχει κάνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυστηρούς κανόνες για τους ε, οίκους αξιολόγησης, για την φερενκιότητα των τραπεζών και για εναντίον των καταχρήσεων. Η Τραπεζική Ένωση είναι λοιπόν κάτι εφικτό. Μπορούμε να το επιτύχουμε πολύ σύντομα εάν εργαστούμε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα υπάρξουν και περαιτέρω προσπάθειες για να εγκρίνουμε την πρωτοβουλία του διπλού πακέτου και για να προωθήσουμε τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσω συνεργασίας. Είναι διαφορετικά, αλλά είναι ουσιότητα δύο αυτά. Μπορούμε να καλέσουμε για περισσότερη ελεγγύη, αν είμαστε δεδεθειμένοι, να δεχτούμε και περισσότερη υπευθυνότητα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ανέφερα μόνο μερικού από του πιο σημαντικού τομεί όπου πρέπει να επικεντρωθούμε του επόμενου μήνε. Φυσικά γνωρίζω το πρόγραμμα τη Κυπριακή Προεδρία είναι πολύ ευρύτερο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε αυτά που μπορούμε να επιτύχουμε σε σχετικά χρονικό διάστημα. Να αναφέρω επίσης και το Σέγγεν και το πακέτο για τα διπλώματα τεχνίας. Ελπίζω ότι και εδώ θα βρούμε καλύτερες λύσεις από αυτές που είναι ενώπιον του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι για να επιτύχει μια Προεδρία του Συμβουλίου χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται αυτή η προσήλωση στους στόχου. Ένα εξάμεινο περνάει πολύ γρήγορα. Χθε, στην συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστόφια και τον πρόεδρο Σούλτ, ανέφερα ότι πρόκειται για τη 17η Προεδρία που θα παρακολουθώ από κοντά. Και σα διαβεβαιώ ότι οι επιτυχημένε Προεδρίε ήταν εκείνε οι οποίε είχαν συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένου στόχου. Να είμαστε ε, παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Η Επιτροπή θα σα βοηθήσει όσο μπορεί για να επιτύχετε και είμαι σίγουρο ότι έτσι θα κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Αρχίζει τώρα η συζήτηση από πλευράς του ΕΛΚΟ Ιώζεφ Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε Χριστόφια, αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια αποφασιστική στιγμή. Το υπενθύμησα και χθες ε, ότι το Συμβούλιο αφιέρωσε 30 συναντήσεις στην οικονομική κρίση και αυτό δεν φτάνει. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την αρχή ενός σχεδίου δράσης. Απαιτείται θάρρος και απαιτείται αποφασιστικότητα και από τη νέα Προεδρία. Μια Προεδρία η οποία θα πείσει ελπίζω τους 26 εταίρους να υπερψηφίσουν μια Ευρώπη ενωμένη, κυρίαρχη γιατί η οικονομική κρίση είναι μια πρόκληση φυσικά, αλλά είναι και μια ευκαιρία, είναι και μια δυνατότητα. Είναι η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και της καταπολέμησης της ανεργίας που έχει φτάσει σε μέσο όρο το 11%. Η ευκαιρία είναι να κάνουμε αυτό το οποίο οι χώρες της Ευρωζώνης έπρεπε να είχαν κάνει εξ αρχής, μια κοινή πολιτική, μια σταθερή πολιτική στον τομέα των δημοσιονομικών και μια πολιτική επενδύσεων μακροπρόθεσμων. Κύριε Πρόεδρε, εμείς είμαστε από δύο εντελώς διαφορετικά αντιτιθέμενα πολιτικά κόμματα. Παρ' όλα αυτά υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες προεδρίας σας. Και κάτι παρατήρησα από αυτά που είπατε και το οποίο μου αρέσει πολύ. Κοινοτική μέθοδος, θα σας στηρίξουμε σε αυτό. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελαν η Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική ε, και να ε, προχωρήσεις με ρυθμούς ανάπτυξης. Πρέπει να δράσουμε γι' αυτό, εποφελούμενοι των 20 γενεθλίων της ενιαίας αγοράς για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που ξεκίνησε ο Ζακ Ντελόρ και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την πράξη για την ενιαία αγορά, να προχωρήσουμε γρήγορα με την οδηγία για τις υπηρεσίες, για την ενιαία ψηφιακή αγορά και να προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε τα βάρη τα οποία υφίστανται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγύηση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση αυτή κύριε Πρόεδρε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Υπάρχει και το θέμα βέβαια της διαπραγμάτευσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας συνειδητοποιώντας ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι ένας επενδυτικός προϋπολογισμός, ένας αναπτυξιακός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός θέσεων απασχόλησης. Το να επενδύσουμε 27 χώρες στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας, της παιδείας, της έρευνας, της καινοτομίας, στι πολιτικές συνοχής, στην διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας των τροφίμων. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα σας στηρίξουμε. Και αυτή είναι μια πραγματική απάντηση στην πρόκληση της κρίσης. Γι' αυτό ακριβώς η Κυπριακή Προεδρία θα βρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν δραστήριο και στρατευμένο συνομιλητή σε σχέση με τις δημοσιονομικές προοπτικές, εφόσον βέβαια ο προϋπολογισμός είναι επαρκής σε σχέση με τις ανάγκες. Θα το ελέγξουμε αυτό, αλλά θα σας βοηθήσουμε να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου με ένα μεγάλο δώρο για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Μη, μη χαμογελάτε κύριε Μπαρόσο, το δώρο δεν θα είναι και για σας. Υπάρχει και κάτι άλλο που ήθελα να πω σήμερα εδώ. Είναι η πολιτική κατάσταση η οποία επικρατεί σε μια χώρα μας στη Ρουμανία εδώ και λίγες μέρες. Η κυρία Ρέντινγκ ήδη εξέφρασε την ζωηρή της ανησυχία. Τι είπε είπε ότι υπήρξαν επιθέσεις ε, εις βάρος της ανεξαρτησίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας από πλευράς της κυβέρνησης. Είπε ότι απαιτείται ένα λειτουργικό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα έτσι ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη στον τομέα της δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Η ομάδα μας συμμερίζεται τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη εγώ την προηγούμενη εβδομάδα εξέφρασα τις ανησυχίες μου σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατικής τάξης στη Ρουμανία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα. Να μην φύγουμε για διακοπές δύο μήνες και τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση αυτή όπως το κάναμε και στο παρελθόν. Μέσα στους επόμενους έξι μήνες θα πρέπει να υπάρξουν βήματα σε όλους αυτούς τους τομείς στους οποίους προανέφερα. Νομίζω ότι έχετε μια μεγάλη δυνατότητα να προσφέρετε στην Ευρώπη κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Άννης Σουόμποντα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση στον συνάδελφο Θα χαιρόμουν αν για την Ουγγαρία είχατε το ίμιση της, ε, των επικρίσεων της κριτικής στάσης ε, που έχετε έναντι της ε, Ρουμανίας. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε χώρα είμαστε υπέρ του ευρωπαϊκού δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών. Πρόεδρε, σας καλοχαιρετίζω με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου που σίγουρα θα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του διότι στεναρά εμπλέκεται. Η Προεδρία σας δεν θα είναι εύκολη Προεδρία. Θα βοηθήσουμε όμως το υποσχόμεθα αυτό για να επιληθούν τα προβλήματα. Εύκολη Προεδρία δεν θα είναι σίγουρα. Η οικονομική κρίση παραμένει ως έχει. Χάνες περίμενε ένα λεπτό λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Δεν υπάρχουν αγγλικά λέτε. Λοιπόν, η αγγλική καμπίνα να μας δώσει ένα μήνυμα αν μπορεί να λειτουργήσει και να διερμηνεύσει. Εντάξει, ωραία, πολύ καλά, ζητώ συγγνώμη, ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή. Παρακαλώ λοιπόν. Λοιπόν, η οικονομική κρίση θα παραμείνει. Η τραπεζική κρίση είναι ισχυρή και εξακολουθεί να υφίσταται. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέστησε σαφέ ότι θα υπάρχει πλήρη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην θέσπιση και δρομολόγηση τη νέα τραπεζική εποπτεία που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτούσαμε. Φυσικά χρειάζονται ειδικοί κανόνε και ρυθμίσει για την Ευρωζώνη, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Κύπρο είναι ένα παράδειγμα. Όποιο δεν είναι στην Ευρωζώνη μπορεί κανεί να το δει αυτό και με την Ελλάδα σε σχέση με τη Ρουμανία αυτό έχει σημαντικότερε επιπτώσει ε, βλαπτική, επιζήμια μορφή, αν δεν είναι κανεί μέρο τη Ευρωζώνη. Και σε σχέση με τι ε, τράπεζε, υπάρχουν πολλοί τραπεζίτε που με τα χρήματα των άλλων ασκούν κερδοσκοπία. Εξακολουθούν πολλοί τραπεζίτε ε, να χειραγωγούν τι αγορέ. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να σταματήσει επιτέλου. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική εποπτεία των τραπεζών στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει του επόμενου μήνε να διασφαλιστεί αποτελεσματικά. Με ιδιαίτερη διαφάνεια για όλε τι τράπεζε. Σε αυτά τα πλαίσια, Πρόεδρε, δύο λόγια για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών πρόσφατα την έκθεση Άνιντ Ποδηματά με μεγάλη πλειοψηφία την εγκρίναμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρω ότι υπάρχουν επιφυλάξει στη χώρα σα, αλλά είναι απόλυτα αναγκαίο να προχωρήσουμε και να θεσπίσουμε τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Δεν θα επιληθούν όλα τα πρόβλημα με αυτό το φόρο, με αυτό το τέλο. Αλλά είπατε ότι πρέπει τα οικονομικά βάρη ισοδίκια να κατανέμονται. Το τέλο χρηματοοικονομική συναλλαγή είναι επιτέλου ένα μέρο, ένα τμήμα τη ισοδίκαια αυτή ε, του ισοδίκαιου επιμερισμού. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε για την αντιμετώπιση και υπέρβαση της κρίσης και μπορεί να συνεισφέρει αυτό και είναι απόλυτα αναγκαίο να συνεισφέρει. Έρχομαι στον προϋπολογισμό, στα δημοσιονομικά. Ο συνάδελφος Ντόλ είπε θα υπάρξει λέει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο με τον προϋπολογισμό του MFF. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό να μην έχουμε, ε, γιορτάσουμε Χριστούγεννα με, μια αρνητική, με ένα αρνητικό συμβιβασμό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που είναι υπέρ του better spending και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι κατά τη συνοχή τη ε, ολοκλήρωση. Τώρα, για τι ε, λιγότερε δαπάνε και σημαντικέ περικοπέ στον προπολογισμό δεν έχετε εμά στο πλευρό σα αν είσαστε υπέρ μια τέτοια θέση. Ε, προσπαθείτε στη Μεγάλη Βρετανία να τα κάνετε αυτά και ε, βλέπετε ποια είναι η αντιμετώπιση σε σχέση με τον πληθυσμό σα. Αν θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο περισσότερη προσπάθεια για τους, τα δημοσιονομικά. Εμεί ως σοσιαλδημοκράτες λέμε ότι θέλουμε και οι περισσότεροι θέλουν να έχουν ένα προϋπολογισμό που θα είναι αποτελεσματικός, να μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματα της ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να υπάρχει και δυνατότητα ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητάς μας. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει κανείς περικοπές και να λέει κάτι περισσότερα για την ανάπτυξη και να περικόπτονται τα κονδύλια. Τα κονδύλια που χρειάζεται κανείς. Όταν ο κύριος Κάμερον στην εκλογική του περιφέρεια χρειάζεται ένα θεσμικό όργανο, πρέπει να το χρηματοδοτήσει όμως σε περιοχές συνοχής, στις περιφέρειες Ένωσης, όπου πρέπει πραγματικά να βοηθήσουμε να προωθηθεί η ανάπτυξη, αν ε, σε σχέση με την αναφορά του Προέδρου είναι στην Πολωνία, Λιθουανία ή σε άλλες χώρες της περιφέρειας, τότε ξαφνικά γίνονται μεγάλε περικοπέ. Και εμεί λέμε όχι, κάθετα σε αυτά, στι περικοπέ αυτέ. Δεν μπορούμε να λέμε χρειαζόμαστε περισσότερε επενδύσει, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και να δίνουμε βάρος, κέντρο βάρους και προσοχή στις περικοπές. Χαίρομαι για το ότι στην Γαλλία υπήρξε μια κίνηση απόκλησης από αυτές τις πολιτικές περικοπών και στην Γερμανία χαίρομαι για το ότι το αναγνώρισε αυτό η κυρία ε, Μέρκελ και σε συζητήσεις με το Σοσιαδημοκρατικό Κόμμα, την S5, ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη πρόθεση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Και θα επιθυμούσα προς αυτό να υπάρξει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, όχι για μας, όχι για το Ευρωκοινοβούλιο, όχι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για του Ευρωπαίου πολίτε που χρειάζονται ένα τέτοιο δώρο με ενδυνάμωση κονδυλίων για την Κυπριακή Προεδρία περνάμε σε μια περιοχή που πλήττεται από μεγάλη κρίση και ισχυρά πλήγματα προσεγγίζουμε την Κύπρο και την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ξέρουμε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση έχει πολύ καλές σχέσεις προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής ε, και ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτές τις σχέσεις πλήρως ε, δεδομένες αυτής της κρίσης. τελευταία παρατήρηση αφορά την Τουρκία. Θλίβομαι και εγώ για ότι η, τη στάση της ε, τουρκικής κυβέρνησης έναντι της Κυπριακής Προεδρίας. Είναι προεδρία της Κυπρι... η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι αν η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα δημιουργούνται προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το όραμα, όραμα της ενιαίας ενωμένης Κύπρου όπου Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι θα μπορούν να ζουν ειρήνη ελληνικά και οι δύο είναι πολίτες της Ευρώπης και πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την, το συνασπισμό των ε, ε, Δημοκρατών και ε, Φιλελευθέρων. Κύριος Βότσον παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η χώρα σας δεν μπορεί να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του μεγέθους της, λόγω της ισχύω της. Οπότε θα πρέπει να ηγηθεί με το σωστό παράδειγμα. Σωστό παράδειγμα στην οικονομική ανάπτυξη. Χρησιμοποιήστε την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση του λαού της Κύπρου. Οικονομολόγοι λένε ότι αυτό θα προσθέσει 12.000 ευρώ στο εισόδημα κάθε οικογένεια στην ίσο σας δώστε το σωστό παράδειγμα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Πάρτε μέτρα εναντίον αυτών των διαφθαρμένων Κυπρίων δικηγόρων και εργολάβων οι οποίοι κλέβουν ε, τις οικονομίες μιας ζωής από τους συνταξιούχους δώστε τα σωστά παραδείγματα, μην παρασυρθείτε από τα τελευταία ευρήματα στον τομέα των υδρογονανθράκων και ξεχάσετε τον ήλιο και τον άνεμο που είναι ο πλούτος της νήσου σας. Μην υποθηκεύσετε τη χώρα σας στη Μόσχα. Μην αποφεύγετε να εμπλακείτε σε συζητήσεις με την Άγκυρα. Προχωρήστε και ε, στις συζητήσεις για τα δημοσιονομικά με τον οδικό χάρτη για το 2050 προσπαθήστε να μειώσετε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ε, θα είστε υπεύθυνοι για τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν για τα δημόσια χρέη και τον έλεγχο των τραπεζών. Χρησιμοποιήστε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης ε, για να βοηθήσετε τις ασθενέστερες χώρες να ανακτήσουν ε, ρυθμούς ανάπτυξης. Να έρθετε σε επαφή με την Τουρκία, να μιλήσετε με την Τουρκία. Μην αγνοείτε το τι υποφέρουν αυτοί που είναι πίσω από το σειρματόπλεγμα του αγκάθωτο μαζί με τους εκλογείς μου από το Γιβλαρτάρ ανήκουν σε αυτούς τους λαούς που έχουν, εξα... που έχουν ξεχαστεί από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται είναι θεματοφύλακες ε, των συνθήκων. Εδώ και 40 χρόνια ένας άλλος νησιώτης από τη Μεσόγειο ο ποιητή τραγουδιστή Ζω Μουστακή μίλησε για τα νησιά, τα γεμάτα αγκαθωτά σηματοπλέγματα που φυλακίζουν τους ανθρώπους του στη Μεσόγειο. Εμείς δεν θα, δεν θα διαμαρτυρηθούμε αν δεν μπορέσετε να φέρετε την ειρήνη και την ελευθερία στη Συρία όσο και αν προσπαθήσετε αλλά παρόλα αυτά προσπαθήστε να διώξετε το σηματόπλεγμα τον αγκαθωτό από το δικό σας το νησί και να προχωρήσετε σε αυτό το οποίο ονομάζει ο ποιητής ένα όμορφο καλοκαίρι που δεν φοβάται το φθινόπωρο. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Βότσον. Ο κύριος Κασουλίδης θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Παρακαλώ κύριε Κασουλίδη. Mr. Watson, don't you think that by addressing this... Κύριε Watson, όταν απευθύνεται μια τέτοια μορφή κριτική σε μια προεδρία που δεν έχει ξεκινήσει καν, είναι κάτι το μη αντικειμενικό, είναι κάτι το μη δίκαιο. Ιδιαίτερα όταν η κριτική αυτή προέρχεται από τη δική σας πλευρά, που αντιπροσωπεύεται μια χώρα η οποία ήταν απεικιοκρατική δύναμη και η οποία έχει ένα τμήμα της ευθύνη για τη διέρεση της συγκεκριμένης νήσου. Με ακριβώς χρησιμοποιώντας τον κανόνα διέρη και βασίλευε. Ε, Παρακαλώ απαντήστε κύριε τώρα. Κύριε Κασουλίδη, εγώ αναγνωρίζω ότι είχε γίνει στα πλαίσια της απεικιοκρατίας από τη χώρα μου. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορηθεί η χώρα μου ότι έχει δημιουργήσει τα προβλήματα της νήσου της Κύπρου. Εγώ δεν κάνω κριτική στην Κύπρο. Χρησιμοποιώ από την Προεδρία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λύσει τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε στην ίσο σα. Αυτό ζητώ. Νομίζω ότι πολλά μένει να γίνουν και εύχομαι στον Πρόεδρο Χριστόφια κάθε επιτυχία προς την κατεύθυνση αυτή και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πρασινών. Η κυρία Ρεμπέκα Χάμς, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ, αφού με τη διάσκεψη των Προέδρων είχαμε πάει στην Κύπρο για την προπαρασκευή της Κυπριακής Προεδρίας, επί μία ημέρα ως ιδιώτης παρέμεινα στη Λευκοσία ώστε να γνωρίσω αυτή την πόλη που δεν γνώριζα. Αφενός στο αρχαιολογικό μουσείο που πήγα και συγκινήθηκα βαθιά πρέπει να πω από την ομορφιά αυτού του, της μεγάλης πολιτιστικής, πολιτισμικής κληρονομιάς της νήσου που γνώρισα εκεί. Και μετά γύρισα στην πραγματικότητα, στην παλαιά πόλη της ε, Λευκοσίας με τα σύνορα, όπου μπορούσε κανείς να περάσει στα σύνορα και πραγματικά συγκλονίστηκα πρέπει να πω από αυτή την αντιπαράθεση, την σύγκρουση που εξακολουθεί και υφίσταται μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Και δεν είμαι τόσο άφρον όπως ο συνάδελφος Γκραμ Γουότσον να σας πω εγώ τι πρέπει να κάνετε για το επόμενο εξάμεινο της Κυπριακής Προεδρίας. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω την επιθυμία που πολλοί από τους συναδέλφους μας σε συζητήσεις στην ε, Λευκοσία ήδη εξέθεσαν ως απόψεις. Η Προεδρία του Συμβουλίου οδηγεί η προσοχή της Ευρώπης να στραφεί στο επίκεντρο της Κύπρου και να συνεισφέρουμε όλοι πρέπει αυτή η πραγματικά αναξιοπρεπής κατάσταση που έχουμε κληρονομήσει από το χθε, από το παρελθόν, να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε, να υπερβούμε αυτή την σύγκρουση, την αντιπαράθεση. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Τούτων λεχθέντων όμως γνωρίζω φυσικά ότι η Προεδρία του Συμβουλίου βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη, δυσχερέστατη κατάσταση αναλαμβάνοντας τη σκητάλη της ε, Προεδρίας. Έχουμε και την αντιπαράθεση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής και δεν ξέρω αν έχουμε ζήσει μια τέτοια Σύνοδο Κορυφής σε περίοδο κρίσης που τα αποτελέσματά της ε, στις αγορές ε, να έχουν τέτοια αποτελέσματα όπως αυτά της ε, τελευταίας συνόδου. Έχουμε επιτόκια που αυξάνονται. Τα επιτόκια για τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυτή την οικονομική κρίση είναι ακόμα υψηλότερα από στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το υπερβούμε. Εσείς αναλαμβάνετε τη σκητάλη της Προεδρίας σε μια χρονική στιγμή που έχει απολύτως λησμονηθεί από πλευράς του Συμβουλίου αυτή η πτυχή όταν γυρνάει κανείς στην πατρίδα του ότι μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή η ευρωπαϊκή κοινότητα μόνο ως κοινότητα αλληλέγγυων υπεύθυνων κρατών μελών. Και από πλευρά των αρχηγών και κρατών κυβερνήσεων και κρατών πρέπει να πούμε ότι κάποιοι από αυτούς είναι περισσότερο κομματικοί κομματική, ε, έχουν κομματική ιδιοτέλεια και δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα της Ευρώπης και την αλληλεγγύη και τα κοινά συμφέροντα. Πρέπει να προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε και μέχρι την χρονική στιγμή όπου η Τρόικα θα συντάξει τη νέα έκθεσή της για την Ελλάδα και για την Κύπρο εξίσου για τη χώρα σας είναι υπαρξιακή αυτή τη στιγμή, υπαρξιακή σπουδαιότητας και σημασίας, ώστε τα προβλήματα από πλευρά του Συμβουλίου μέχρι τότε να έχουν ξεπεραστεί. Εγώ τουλάχιστον από πλευρά μου ανησυχώ ιδιαίτερα για την επιρροή αυτή της νέας έκθεσης της Τρόικας για την Ελλάδα που αναμένεται για να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ θα έλεγα ε, ευαίσθητη περιοχή, ευάλωτο είναι το θέμα, ευαίσθητο και πρέπει να δούμε και αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει νομίζω θετικούς προσανατολισμούς για αυτά που κατεπηγόντως χρειάζονται και πρέπει να ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια αυτού του θέρους. Θα ήθελα να τα αναφέρω αυτά και να σας τα πω κύριε Χριστόφια γιατί πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, το δίκαιο είναι κάτι στο οποίο ιδιαίτερα καταβάλλετε προσπάθειες και είναι μέσα στην ψυχή σας. Και γνωρίζω πως έχουν τα διαθωτικά προβλήματα με τις μεγάλες τράπεζες και τον χρηματοοικονομικό τομέα και στην Κύπρο πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ε, για την φορολογική δικαιοσύνη. Να αντιμετωπιστούν ε, οι φορολογικές οάσεις, ε, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή. Την δική σας προεδρία θα μπορέσετε να την οδηγήσετε σε αίσιο πέρας μόνο όταν αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα προβλήματα και είσαστε επιτυχεί. Σα ευχαριστώ κυρία Χάρμ. Στη συνέχεια για του Ευρωπαίου Συντηρητικού θα λέει τον λόγο Ευρωβουλευτή κ. Κάλαχαν, παρακαλώ. All... Καταρχά, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Χριστόφια για την ε, παρουσίασή του και για την, ε, το καλωσόρισμα που ε, έκανε στην ομάδα μας όταν πρόσφατα επισκεφθήκαμε την Κύπρο. Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τις επικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε με εκείνον και την κυβέρνησή του. Τώρα βεβαίως είναι σαφές ότι δεν έχουμε πολλά κοινά σημεία από πλευρά πολιτική, αλλά εκτιμούμε ιδιαίτερα την ε, ευγένεια και φιλοξενία του και συμφωνούμε με, τις, ε, ε, με αυτό που είπε στην ομιλία του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μοιάζει να αφορά πολλούς Ευρωπαίους πολίτες πρέπει να γίνει πολύ πιο έντονη η παρουσία της η θέση μας είναι σαφής δεν θέλουμε να αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αν συνεχίσει να ακολουθεί τα θέματα του παρελθόντος την ημέρηση διάταξη του παρελθόντος οπωσδήποτε θα αποτύχει και να πω κάτι και στον πρόεδρο Μπαρόσο. Με εξέπληξε ιδιαίτερα η έκρηξή του χθε εδώ στην Ολομέλεια όπου ε, έμοιαζε να λέει ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι το ευρώ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Αυτά είναι παράλογα. Πιστεύουμε Εντελώ άλλα πράγματα. Εκείνο που μα ανησυχεί είναι ότι πολλοί άνθρωποι υποφέρουν λόγω των πολιτικών σα επιλογών. Έχω αναφέρει πολύ συχνά ποιε νομίζω είναι εναλλακτικέ λύσει για το ευρώ ή μια αποτελεσματική δημοσιονομική ένωση ή μια μείωση στο μέγεθο τη ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή προσπαθείτε να οδεύσετε προ μια πολιτική ένωση χωρί τη δημοσιονομική ένωση που είναι προπόθεση. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για το τι θα σημαίνει αυτό για, τις, ε, για τη δημοκρατία σε πολλές χώρες μέλη. Αν θα είτε επιζήσει είτε δεν επιζήσει το ευρώ, νομίζω ότι οι χώρες που είχαν ε, την κοινή λογική να μην ενταχθούν δεν είναι υποχρεωμένες να οδεύσουν ε, προς περισσότερη ενοποίηση εάν δεν το επιθυμούν. Αλλά ένα όργανο πρέπει οπωσδήποτε να είναι κοινή διοκτησία για των 27 χωρών είναι η αγορά είναι ένα στοιχείο που όλοι υποστηρίζουμε και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κυπριακή Προεδρία τόνισε ότι μία από τις φιλοδοξίες της είναι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Θα έχετε την πλήρη στήριξή μας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η Προεδρία θα καταλήξει τις ε, διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τις ε, κεφαλικές ανάγκες. Ε, χθες ο πρόεδρος Μπαρόσο τόνισε ότι οι προηγούμενε ουσιαστικέ κυβερνήσει του Ηνωμένου Βασιλείου ε, έδωσαν πολλά δισεκατομμύρια στι τράπεζε για να επιβιώσουν. Ε, είναι στόχο μα φυσικά να, έχει, να έχουν επαρκέ κεφάλαιο τράπεζε ώστε να μην ξαναχρειαστεί αυτή η διάσωση των τραπεζών. Γιατί προσπαθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τι ε, προσπάθειε που έκανε στη Βασιλεία το Ηνωμένο Βασίλειο για να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία για την κεφαλαιοποίηση. Εμεί θα πρέπει να είμαστε γιατί εμείς ως κράτος είμαστε πολύ πιο αυστηροί από ό,τι είστε εσείς για τις ε, προϋποθέσεις για τις τράπεζες. Θέλουμε οπωσδήποτε να μην χρειαστεί διάσωση των τραπεζών. Και να περάσω στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εξακολουθεί να με εκπλήσει το πώς η Κομισιόν θα μπορέσει να εφαρμόσει λιτότητα στα κράτη-μέλη, ενώ παράλληλα απαιτεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη περισσότερα χρήματα για τον κοινοτικό προπολογισμό. Όλοι πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσει, φαίνεται, εκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πετάμε χρήματα λοιπόν στα οικονομικά προβλήματα, νομίζουμε ότι έτσι θα τα λύσουμε. Πρόκειται για ένα δόγμα το οποίο στη δεκαετία του 70 καταδείχθηκε ω ανεπαρκέ. Και αν ε, θα μα υποβάλλετε έναν προπολογισμό που θα έχει ποιοτικού στόχου καλύτερη δαπάνη των χρημάτων, όχι περισσότερα χρήματα, τότε οπωσδήποτε θα σα υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κάλαναν για ε, την ε, Νέα Ευρωπαϊκή Αριστερά, η κυρία Τσίμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αξιότιμη κύριε Δημήτρη Χριστόφια, για μένα είναι σήμερα και για την κοινοβουλευτική μου ομάδα ιδιαίτερα σημαντική στιγμή να σας καλωσορίζω και να σας προσφωνήσω ως Προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε επίσης ιδιαίτερα διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας άνθρωπος που ανήκει στην δική μας πολιτική οικογένεια. Αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια χρονική συγκυρία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και πρέπει να θέσουμε την τροχιά και την πορεία και να δούμε αν πραγματικά θα τα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν, και αυτό πιστεύω εγώ ότι θα ήταν μια ιστορική ήττα, θα γίνει μόνο μια υποσημείωση τη ιστορία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω από συζητήσει που είχαμε μαζί σα και με του εκπροσώπου τη κυβέρνησή σα και με του προέδρου των κοινοβουλευτικών ομάδων, πολιτικών ομάδων και κομμάτων στη χώρα σα ότι έχουν προετοιμαστεί εξαιρετικά για τη δική σας Προεδρία όλοι. Και σε αυτή την εμβέλεια, σε αυτό το εύρος, σε αυτό το φάρμα, συγγνώμη, έχουν προετοιμαστεί και είναι ικανοί να προχωρήσουν. Όμως αποσαφηνίστηκε ότι θέλετε συνειδητά να στρέψετε την προσοχή των κυβερνώντων στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Και μπορώ να σα πω μετά από όλα όσα άκουσα τα τελευταία χρόνια, είναι η πρώτη φορά που ένα προεδρεύων τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακριβώ αυτό το προαναγγέλει και το κάνει και λέει αυτό και εγώ είδα ότι αυτό έλειπε από τους ε, επίσημους λόγους που ε, το Δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής μας. Εκείνοι που υφίστανται τα μεγαλύτερα βάρη και πλήγματα. Θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί αυτό, αλλά πολλά θα είχαμε κερδίσει και θα ήταν θετικό αυτό. Και είμαι βέβαια ότι θα προχωρήσετε και θα τα κάνετε αυτά, αν θα δώσετε το θάρρος στους ανθρώπους, τους ενθαρρύνετε με την Προεδρία σας να προσπαθήσετε να καταβάλλετε προσπάθειες υπέρ των δικαιωμάτων τους και να συνεισφέρετε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνειδητοποιήσουν αυτά τα προβλήματα. Πάντα κάνουμε λόγο για το ευρώ και την νομισματική σταθερότητα, ανάγκη που και εγώ αναγνωρίζω ότι υφίσταται και που είναι σημαντική υπόθεση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο. Υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις και όροι που έχουν καθοριστεί. Δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός και στόχος, αυτός το, αυτονόητος αποκλειστικά στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσουν όλα αυτά και να πεινάνε οι άνθρωποι και να καταρρεύσουν τα κοινωνικά συστήματα και να μην έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Εδώ έχουν αντιστραφεί οι όροι. Δεν είναι αυτό που εμεί ε, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε στόχο και νόημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα υποστηρίζουμε λοιπόν έντονα και στεναρά στην προσπάθειά σα να υπάρξει αλληλεγγύη σε σχέση με τα κράτη-μέλη, μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ε, κοινωνικών ομάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορέσει να όχι να δρά ω ε, υπέρμαχο μια μικρή ομάδα ομάδας κοινωνικής ομάδας ε, ή πληθυσμιακής ομάδα, αλλά υπέρ του συνόλου των πολιτών. Και θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο να κάνω για να υπογραμμίσω ότι όλα αυτά που εσείς αναφέρατε και απαριθμίσατε ως προτεραιότητες είναι πολύ σημαντικά και για μας και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να πορευτούμε όπως το σκιαγραφίσατε εσείς. Κάντε όμως κάτι κι εσείς παρακαλώ επιτέλους ώστε να μην φοβούνται πια οι πολίτες. Να μην φοβούνται. Ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος για τις δημοκρατίες. Και πιστεύω ότι κάποιες από τις αποφάσεις τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ιδιαίτερα στις εκλογές στην Ελλάδα και σε σχέση με την, ε, το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία χαρακτηρίστηκαν από φοβίε και φόβου. Και αν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουμε να υπάρχουν φοβίε και φόβοι για του πολίτε και έτσι να λαμβάνουν αποφάσει, αυτό δεν είναι καλό σύμβουλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσίμερ για την ομάδα EFD, η κυρία Σαβέλα. Κύριε Πρόεδρε Χριστόφια, σας καλωσορίζουμε στην Προεδρία και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία η κυπριακή προεδρία ξεκινάει εν μέσω μεγάλων πολιτικών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή ένωση. μετά τις αποφάσεις του συμβουλίου του ιουλίου κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας πρέπει να προωθηθούν η οικονομική τραπεζική και πολιτική ενοποίηση της ευρώπης. κυρίες και κύριοι αυτό το οποίο ίσως δεν ξέρετε είναι ότι αυτή η μικρή χώρα η κύπρος χαρακτηρίζεται από ανθρώπους που έχουν ορθολογισμό, πειθαρχία και τόλμη. Η Κύπρος βλέποντας πώς προχώρησε το γειτονικό της Ισραήλ στην επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας με την εξέβρεση φυσικού αερίου προχώρησαν τολμηρά και ορθολογικά σε μια συμμαχία επιχειρηματική με το Ισραήλ χωρίς να διαταράξουν τις σχέσεις τους με τον αραβικό κόσμο προσβλέποντας σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους εμάς να δούμε πώς ο τομέας της ενέργειας μπορεί να μεταβληθεί και να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας. επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει όπως ετονίστηκε νωρίτερα να αξιοποιήσουμε τις καλές σχέσεις της κυπριακής δημοκρατίας με πάρα πολλές χώρες του τρίτου κόσμου ιδιαίτερα με τον αραβικό κόσμο. καλή επιτυχία κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Τζαβέλα. Ε, από πλευρά των μη εγγεγραμμένων η κυρία Σινκλέα. Ε, ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Με χαρά σας συνάντησα όταν ε, ήρθα το 2009 στη Λευκοσία και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στην προσπάθεια που κάνετε για να επιλύσετε το Κυπριακό. Ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να έχει επιλυθεί εδώ και καιρό και ελπίζω η προσβολή που σας έκανε ως Προεδρία η τουρκική κυβέρνηση το ότι δεν σας αναγνώρισε ως Πρόεδρο της Κύπρου αυτό θα πρέπει να τονιστεί εδώ μέσα. θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει ή να αφαιρέσει το καθεστώ τη υποψήφια χώρα από την Τουρκία γιατί δεν είναι διατεθειμένοι να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι είναι προπήριο δημοκρατίας. Αλλά εκπαιδευθήκατε στη Ρωσία. Θα είδατε πως η Ντούμα δεν ήταν προπύργιο δημοκρατία ε, περισσότερο από εδώ. Και το Πολίτμπυρο ε, της Σοβιετικής Ένωσης μπορεί να συγκριθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τονίσατε τι προβλήματα έχει η Προεδρία σας. Ε, τονίσατε ε, τα δεινά των εργαζομένων. Στην Αθήνα υπάρχουν επιγραφές ε, στους τοίχους που λένε να μην ζήσουμε ως σκλάβοι. Αλλά η ιδεολογία σας ως κομμουνιστή θα κάνει πολύ δύσκολο να επιτύχετε αυτούς τους στόχους. Πώς θα προστατεύσετε τους εργαζόμενους, τους εργάτες μέσω της λιτότητας που επιβάλλει η Άγγελα Μέρκελ και η λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 δεν έχει κανένα όραμα το 2020. Θα επιτύχει αναμφίβολα κατά τη γνώμη μου όπως και η στρατηγική της Λισαβόνας που είχε στόχο το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ανταγωνιστική και βασισμένη σε γνώση ε, οικονομία. Είπατε ότι δεν πρέπει να περιμένετε τρομερά επιτεύγματα, ένα βουνό ολόκληρο από την ε, Κύπρο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το έβερε των ε, προσδοκιών όλων. Ευχαριστώ. Από πλευρά ΕΛΚ, ο κύριο Κασουλίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία με αποφασιστικότητα και ταπεινότητα, έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του θεσμού έχετε αναπτύξει κύριε πρόεδρε της κυπριακής δημοκρατίας τις προτεραιότητες της προεδρίας σας το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο το κοινό άσυλο την πολιτική της προώθησης του κεφαλαίου της ε, αγροτικής πολιτικής την ενιαία ναυτιλιακή πολιτική την ενέργεια κλπ. η προγραμματιζόμενη σύνοδος των υπουργών εξωτερικών των κρατών μελών της ένωσης και του αραβικού συνδέσμου μαρτυρεί το μεγάλο ενδιαφέρον για τις χώρες της αραβικής άνοιξης. η προεδρία σας ασφαλώς θα προχωρήσει και το θέμα της διεύρυνσης περιλαμβανομένης και της τουρκίας την οποία είμαι σίγουρος ότι θα χειριστείτε με αμεροληψία και δίκαια. λυπούμαστε για τη στάση της τουρκίας απέναντι στην προεδρία δεν σέβεται τους θεσμούς διότι η προεδρία είναι θεσμός της ένωσης και για έξι μήνες δεν είναι η χώρα με τις διμερείς διαφορές που τυχόν η τουρκία να έχει. η παράδοση θέλει την εκάστοτε προεδρία να αφήνει κατά μέρο τα δικά της εθνικά προβλήματα και να αφοσιώνεται στα προβλήματα της ευρώπης και αυτόν έχετε δηλώσει ότι πρόκειται να πράξετε. έστω και αν η τουρκία με τις απειλές που εκτοξεύει εις βάρος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θέλει να αποσπάσει την προσοχή από τους στόχους της προεδρίας. η κύπρος καλείται να αποδείξει ότι με την προεδρία της αποτελεί ένα σοβαρό και αξιόπιστο εταίρο. ταυτόχρονα όμως η επιτυχία της θα είναι η απάντηση σε δηλώσεις από τους κυρίους ερντογάν και Μπαγής που έγιναν και αναφέρω ότι δεν είμαστε καν κράτος είμαστε μισό κράτος ούτε καν φιλή προεδρεύουσα μιας μίζερης ευρώπης δηλώσεις δικές τους. δυστυχώς η έναρξη της προεδρίας συμπίπτει με την προθεσμία κεφαλαιοποίησης των τραπεζών όλης της ευρώπης. αυτό μας οδηγεί στον μηχανισμό στήριξης Όμω η οικονομία τη κύπρου καταστράφηκε το 1974 από την τουρκική εισβολή και η εργατικότητα του κυπριακού λαού δημιούργησε έναν οικονομικό θαύμα. αυτό θα πράξει ξανά στα προσεχή χρόνια. σας ευχαριστώ. Η κυρία Σινκλέρ, θέλετε να κάνετε μια ερώτηση στον κύριο Κασουλίδη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κασουλίδη γιατί θεωρεί ότι η επίθεση ήταν αιτιολογημένη στον Ηνωμένο Βασίλειο. Η χώρα μου έχει δώσει δέκα δις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χώρα του και οι δυνάμεις μας είναι εκεί για να σας υπερασπιστούν και εξοδεύουν πολλά χρήματα. Εάν δεν ήταν οι δυνάμεις μας εκεί η Τουρκία θα είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο το 1974. Αλλά γιατί να μιλάμε για το παρελθόν, να μιλήσουμε για τον Ιταλικό, την Ιταλική επικοινοκρατία, την Πορτογαλική, για την Αυστρο-Ουγγαρία, για την Γερμανική επικρατικότητα. Θα μιλήσουμε για το παρελθόν ή για το μέλλον. Θέλετε να είστε μέλο του τμήμα του παρελθόντο. Παρακαλώ κύριε Κασουλίδη λόγω της παρουσίας των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, η σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου πρέπει να είναι και είναι άριστες. Και ελπίζω τα σχόλια αυτά που έρχονται από εκπροσώπους του Βρετανικού λαού θα έπρεπε επίσης να μην ασχολούνται με τον παρελθόν, να μην θυμίζουν την πολιτική διέρη και βασίλευε που οδήγησαν στην ε, ε, διαίρεση της Κύπρου για την οποία φέρουν τμήμα της ευθύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από πλευρά Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ο κύριος Μαυρονικόλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Χριστόφια σε σχέση με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει για την εξάμηνη Προεδρία της Κύπρου είναι μια τοποθέτηση η οποία είναι προοδευτική αναδεικνύει τα σημαντικά προβλήματα της ένωσης και ιδιαίτερα την μεγάλη οικονομική κρίση και την αντιμετωπίζει με έναν προοδευτικό και δημοκρατικό τρόπο που αυτό σημαίνει εν ολίγης ότι δεν αποδέχεται ως μοναδική έξοδο από την οικονομική κρίση την πολιτική της αυστηρής λιτότητας αλλά παράλληλα μιλά για καταπολέμηση της ανεργίας για αξιοποίηση της ανάπτυξης και για τη δημιουργία ενός νέου πλέγματος εντός της ένωσης που πραγματικά να δίνει ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη και έξοδο από την ύφεση. δεύτερον αναδεικνύει σεβασμό απέναντι στις αρχές της ευρωπαϊκής ένωσης για ισότητα δημοκρατία αλληλεγγύη κοινωνική συνοχή αυτές οι ίδιες αρχές οι οποίες φέρουν σήμερα εδώ τον πρόεδρο της κυπριακής δημοκρατίας ως πρόεδρο ολόκληρης της ευρωπαϊκής ένωσης. άρα αγωνιζόμαστε όλοι μας για να αναπτύξουμε την δική μας οικογένεια. αγωνιζόμαστε όλοι μας για περισσότερη ευρώπη και αυτό είναι το στίγμα της πολιτικής που ανέπτυξε ο πρόεδρος της κυπριακής δημοκρατίας. ορθά ο πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο πρόβλημα του νησιού στο κυπριακό πρόβλημα. είναι όμως γεγονός ότι οι δεκάδες ή εκατοντάδες ακόμα επισκέψεις ευρωβουλευτών σήμερα στην κυπριακή δημοκρατία βλέπουν τις πραγματικότητες βλέπουν την διχασμένη πρωτεύουσα τη λευκοσία την μοναδική διχασμένη πρωτεύουσα παγκοσμίω βλέπουν την ισχυρή τουρκική κατοχική παρουσία 45.000 τουρκικός κατοχικός στρατός για να προστατεύσει δήθεν και σε εισαγωγικά μια τουρκοκυπριακή κοινότητα των εκατό χιλιάδων ατόμων. Αγωνιούμε εμείς περισσότερον από όλους για την τουρκοκυπριακή κοινότητα διότι μέσω αυτής πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. αντίθετα η τουρκία η οποία δεν αναγνωρίζει την κυπριακή δημοκρατία δεν αναγνωρίζει σήμερα που μιλούμε την προεδρία της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης με το μόνο πράγμα που ασχολείται είναι με τον σταδιακό επικισμό του νησιού και την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού. 700.000 έπικοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα και θα είναι παράδοξο και είναι παράδοξο να υπάρχουν βουλευτές ή και αρχηγοί πολιτικών ομάδων όπως ο κύριος Βάτσον οι οποίοι να αντιμετωπίζουν το κυπριακό πρόβλημα λες και το δημιούργησαν οι κύπροι. τελειώνω με μια ακαδημαϊκή ερώτηση θα συνεχίσει απρόσκοπτα η ενταξιακή πορεία της τουρκίας κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους τώρα το λόγο η κυρία σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στα ελληνικά κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να αναφέρω το ότι τώρα σήμερα έχουμε ένα ισορροπημένο ευφυές πρόγραμμα της Προεδρίας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εφαρμογή, στην υλοποίηση του. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν υποσχεθεί στους Ευρωπαίους πολίτες ότι θα υπάρξει ένα κοινό κοινοτικό σύστημα το οποίο θα δημιουργηθεί πριν από τα τέλη του έτους και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση τώρα που αντιμετωπίζει και η Κυπριακή Προεδρία, η Κύπρος. Όλα βρίσκονται τώρα στα χέρια της Κύπρου. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, τεράστια εμπιστοσύνη στις ικανότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. όμως ωστόσο όλα αυτά, πρέπει να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μα. Και μάλιστα άμεσα. Όσον αφορά τη Συμφωνία Δουβλίνου 2, είμαστε Είμαι συγγήτρια και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια απόφαση. Θα ήθελα να συζητήσω όμως, να ζητήσω να ενδυναμώσετε τις προσπάθειές σας σε αυτό το διάστημα, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε, να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε στους πολίτες μας. Και σε άλλους ε, θεματικούς τομείς ε, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα, το ευρωπαϊκό δίπλωμα Τεχνίας. Μία πιθανή μας χωρίζει μόνο από την ε, συμφωνία. Επί δεκαετίες ε, διαπραγματευόμαστε. Τώρα μπορούμε στους εφευρέτες να προσφέρουμε ένα ενιαίο δίπλωμα ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας. Το κόστος, οι δαπάνες ε, θα μειωθούν. Και πρέπει να είμαστε ευφυείς στον τρόπο, εφάνταστοι στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε και με σθένος. Έτσι πρέπει να διαπραγματευτούμε και να προχωρήσουμε. Αν καταφέρει η Κυπριακή Προεδρία Κύπρος να υλοποιήσει αυτές τις προκλήσεις και να αντιμετωπίσει αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει και να πετύχει αυτού του στόχου, τότε θα θυμόμαστε ότι είναι με μια μικρή χώρα, αλλά με μεγάλη σπουδαιότητα και που ιδιαίτερα σημαντικά συνεισέφερε για την επίτευξη των στόχων τη Προεδρία. Σα ευχαριστώ, σα εύχομαι κάθε επιτυχία με τι προσπάθειέ Είναι Φιλίπ Λομπέρ. Φιλίπ Λομπέρ, παρακαλώ, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε κύριε Πρόεδρε. Θα σας επευθύνω το λόγο σαν εκπρόσωπο μίας από τις 27 χώρες. Ακούγοντάς σας και μετά από τον κύριο Βαν και βλέποντας τις δράσεις του Συμβουλίου έχω την εντύπωση ότι εδώ έχουμε μια, ένα διχασμό προσωπικότητα στην καλύτερη περίπτωση για να μην πω κάτι περισσότερο. Λέει από τη μία το Συμβουλίο θέλουμε δημοσιονομική Ένωση και από την άλλη είναι κατά ενός σοβαρού προϋπολογισμού με πραγματικούς ιδίους πόρους για να τον μεταχειρίζεται και να τον χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά λέει το Συμβούλιο θέλουμε δημοσιονομική ένωση. Δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να μην καταπολεμά συστηματικά σύμφωνα με το δόγμα εναντίωσης της εναρμόνισης της φορολογικής. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είδα ότι το Συμβούλιο αρνήθηκε κατηγορηματικά οι εσδήποτε ε, μορφές περιορισμού για τα venture capital τα οποία ε, προσφεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες είναι φορολογική παράδοση ή φιλοξενούν φορολογικούς παραδείσους. Ίσως αυτό κάτι να εξηγεί. Χρειάζεται εδώ να υπάρχει μεγαλύτερη εν πάση περιπτώσει ε, μορφή ελέγχου δημοκρατικού. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όλοι εσείς λέτε καλά λόγια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά όταν αναλαμβάνετε δράση, κάθε δράση σας προσπαθεί να αγνοήσει και ε, να βγάλει από τη μέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν συζητάμε τα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης κάνετε ένα δημοσιονομικό σύμφωνο το οποίο αγνοεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν μιλάμε για την Τραπεζική Ένωση το κάνετε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην λάβετε υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν ποιο είναι το πρόσωπο του Συμβουλίου τους επόμενους έξι μήνες. Είναι το του Δόκτωρος Τζέκιλ ή αυτό του κ. Χάιντ. Ευχαριστώ για από πλευρά τη ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριο Ζαχραντήλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Χριστόφια. Οι χώρε μα ταυτόχρονα εντάχθηκαν, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό τον λόγο χαίρομαι ιδιαίτερα εγώ σήμερα για το ότι ένα περαιτέρω νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα αναλαμβάνει τη σκητάλη της Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μπορεί να είναι μικρή η Κύπρος. Εμείς επισκεφθήκαμε πρόσφατα την Κύπρο, σας συναντήσαμε, συναντήσαμε τους υπουργούς της κυβέρνησής μας, ε, την Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Εξωτερικών και όλα αυτά δημιούργησαν και άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Έχετε προετοιμαστεί εξαιρετικά για την Προεδρία σας. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα αυτής της επίσκεψης ημών στη χώρα σας, για τον τρόπο με τον οποίο μας υποδεχθήκατε, μας καλοδεχθήκατε και διαβουλευθήκατε μαζί, σας, μαζί μας. Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν επιφυλάξεις, ε, μακάρι να ήταν οι καλύτερες λύσεις αυτές. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι ένα θετικό βήμα αυτό και δεν συμφωνώ με τον κύριο Μπαρόζο και δυστυχώς δεν συμφωνώ και η πλειοψηφία σε σχέση με την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πιστεύει ότι είναι μια καλή πρόταση για λύση αυτή. Κάνατε λόγο για την αρχή της αλληλεγγύης. Εδώ πρέπει να προσέξουμε όμως αυτή η αρχή να μην οδηγήσει στο ότι θα γίνει μια ένωση μετάθεση κονδυλίων και μεταφορά κονδυλίων από τη μια χώρα στην άλλη. Αποκλειστικά και μόνο αυτό. Αυτό θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες εντάσεις ε, μεταξύ των διαφορετικών λαών. Και σε σχέση με τις προκατακτικέ δράσεις για ένα νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χρηματοδοτικό πλαίσιο, πολιτέ πλαίσιο για το οποίο θα είσαστε αρμόδιο ε, ο ρεαλισμό και η πραγματιστική προσέγγιση όπω ε, από εσά διαγραφήθηκαν σε σχέση με τα φορολογικά θέματα ή σε σχέση με τις ρυθμίσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, στις προσπάθειές σας αυτές ε, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μας. Δεν χρειαζόμαστε ένα τέλος ε, ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Θέλουμε τον ανταγωνισμό να τον διασφαλίσουμε αποτελεσματικά ώστε να είναι λειτουργική η Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και ελπίζω ότι θα στεφθεί με επιτυχία η Προεδρία σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου παρακαλώ. Καλημέρα σα. Καλωσορίζω και εγώ καταρχήν τον Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Κύπρος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα μικρό κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έκταση μερικέ δεκάδε φορέ μικρότερη από σχεδόν κάθε άλλο κράτο τη Ένωση. Με πληθυσμό που ισοδυναμεί με το 1 τέταρτο των πολιτών του Βερολίνου και το 1 δέκατο, αν δεν κάνω λάθο, αυτών του Λονδίνου ταυτόχρονα είναι ένα κράτο του οποίου το ένα τρίτο των εδαφών του κατέχεται από χώρα που αναζητά την ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση. μόνο όμω αν ένα τέτοιο κράτο στηριχτεί ομόθυμα από τα υπόλοιπα 26 κράτη και από όλου εσά του συνάδελφου ευρωβουλευτέ. μόνο έτσι μπορεί να αποδειχθεί ότι η ένωση αντιλαμβάνεται τον εαυτό τη ω αμφικτιονία ισοτήμων και αλληλέγγυων κρατών και πολιτών η κύπρος μικρή χώρα υπό ημικατοχή χρειάζεται τη δική μας ασπίδα προστασίας ως ευρωκοινοβούλιο. καλούμε την ευρωπαϊκή ένωση να απαντήσει επίσημα και καθαρά στην τουρκία η οποία δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι δεν θα έχει καμία επαφή με την κυπριακή προεδρία και η μόνη απάντηση είναι πως η επιτροπή και το συμβούλιο δεν πρέπει αυτοί να έχουν καμία επαφή με την τουρκία ενώ η χώρα αυτή δεν αναγνωρίζει την προεδρία της ένωσης σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι βιώνουμε μια κρίση που κυριολεκτικά πίνει το αίμα των οικοκυριών. υπάρχει ασυδοσία των λεγόμενων αγορών και η παντελής έλλειψη εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα οδηγούν σε αύξηση του δημοσίου χρέους στέλνοντας τους εργαζόμενους στην ένδια και τον εξευτελισμό. καλούμε το ευρωκοινοβούλιο και την ένωση να στηρίξει τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας και το κοινωνικό της μήνυμα για την εξάλληψη της φτώχεια και ειδικότερα της παιδικής την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή της μεσογείου καθώς και την ολοκλήρωση της ενιαίας πολιτικής ασύλου. Ευχαριστώ. Τώρα από πλευρά τη ομάδα ε, τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία, ε, Ο κύριο Μοργάντη. Θα ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερα στην Κυπριακή Προεδρία η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο πολιτικό. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι από πλευράς μου και από πλευράς του κόμματός μου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τουρκικές πιέσεις όπως το κάναμε στο παρελθόν. Η Ευρώπη κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην Κύπρο. Εγώ σας επισκέφτηκα εδώ και λίγους μήνες και μπόρεσα να διαπιστώσω η διεισόμαση ε, πραγματικά τη βλάβη, τις ζημίες τις οποίες προκάλεσαν σε επίπεδο πολιτιστικό, σε επίπεδο κληρονομιάς ε, οι Τούρκοι στο βόρειο τμήμα του νησιού. Η Ευρώπη από το 2007 μέχρι το 2013 έδωσε 5 δις στην Τουρκία, μια χώρα με οικονομική ανάπτυξη ισχυρή. Και πέρυσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσε στην Τουρκία πάνω από 2 δις δάνεια. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα να σκέφτεται τις δικές της χώρες και να μην βοηθάει αυτές τις χώρες οι οποίες απειλούν τις χώρες της Ένωσης. Η κυρία Βέρτμαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας στα ελληνικά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαίρουμε τον πρόεδρο Χριστόφια και την ομάδα του για την εξαιρετική προετοιμασία της Κύπρου για την Προεδρία στην ιστορία αυτό είναι ένα ορόσημο. Μία από τι πιο μικρέ, νεότερε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση επομίζεται μια τέτοια τεράστια πρόκληση σε πολύ δυσχερή οικονομική συγκυρία και περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο τμήματα του προγράμματό σα έχουν τεράστια σημασία. Η επικέντρωση στα συμφέροντα των πολιτών και το ε, MFF το Multi-Annual Financial Framework, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παγκόσμια και όσον αφορά την απήχηση σε σχέση με την Κύπρο και την Προεδρία της από την, τον τουρκικό ε, τύπο πρέπει να είναι ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ομιλεί με μια φωνή. Πρέπει όλα τα ψηφίσματα να εφαρμοστούν και όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνουν σεβαστοί και σεβαστά από όλους και από την Τουρκία. Ας εργαστούμε λοιπόν όλοι παρακαλώ και ας υποστηρίξουμε την Προεδρία της Ένωσης ε, την Κύπρο. Σας ευχαριστώ στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ στη συνέχεια εξ ονόματος του Έλκο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε για την προετοίμαση, για τους επόμενους έξι μήνες που θα είναι τεράστια σπουδαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομίζεστε τεράστιες ευθύνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά της χώρας σας, της Κύπρου και αναμένουμε ότι θα έχουμε κατά το τέλη του 2012 ένα θετικό ισολογισμό. Τα πιο σημαντικά θέματα είναι οι οριζόντιες εγκάρσεις πολιτικές και το MFF και από πλευράς Δανέζικης Προεδρίας δεν έχετε κληροδότημα πλούσιο σε σχέση με αυτά. Για τον προπολογισμό, για τα δημοσιονομικά θέματα, δημοσιονομικά θέματα δεν αναφέρθηκε ούτε λέξη, ενώ αυτά είναι τα πιο σημαντικά και για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης ασχολήθηκε η Προεδρία αυτή για ε, θέματα της, ε, ε, των οριζόντιων πολιτικών υπό την συναπόφαση. Τώρα είναι έργο της δικής σας Προεδρίας που ακολουθεί η συζήτηση με το Ευρωκοινοβούλιο να ξαναξεκινήσει και να ενδυναμωθεί ώστε να έχουμε ένα προϋπολογισμό που θα συμφωνηθεί εφέτος και θα είναι αποτελεσματικός. Έχετε διαμεσολαβητικό ρόλο ως προς αυτά στον τομέα μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά και τα θέματα Σέγγεν τα κράτη-μέλη εκείνα που έχουν εξωτερικά σύνορα ζητούν να μην υπάρξουν περικοπές όσον αφορά τα κονδύλια για τις ε, δράσεις ε, Σέγγεν και να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με άλλες χώρες. Έχετε το έργο το οποίο ε, επομίζεστε. Πρέπει να προσπαθήσετε να επιλύσετε όλα αυτά τα προβλήματα επιτυχώς. Και αναφέρθηκε το θέμα της Ουγγαρίας από τον κύριο Σβόβοντα όταν γίνεται λόγος για τη Ρουμανία. Είναι πρόεδρος μιας μεγάλης κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου και πρέπει να γνωρίζει τι σημαίνουν οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και ποια σημασία έχουν στην Ρουμανία, Ουγγαρία και στην Αυστρία. Στην Ρουμανία δεν υπάρχει σε σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση κάτι το ε, διαφορετικό. Βλέπει κανείς μια επίθεση κατά της δημοκρατίας. Υπάρχουν ε, θέματα του προσφυγών στο συνταγματικό δικαστήριο. Υπάρχουν, ε, υπάρχει παραβίαση ή περιφρόνηση έναντι σημαντικών αρχών και δικαστηρίων και αυτά είναι σημαντικές επεμβάσεις ή παρεμβάσεις στις βάρος της δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν καταβάλουμε προσπάθειες για την προάσπιση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Για τη σοσιαλιστική ομάδα κύριο Σκοφεράτη, Κοφεράτη παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας περιμένει ένα δύσκολο εξάμεινο, αλλά υπάρχει μια προτεραιότητα απόλυτη και η προτεραιότητα αυτή ονομάζεται ανάπτυξη. Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι χρήσιμη, είναι σημαντική, αφεαυτής όμω δεν δίνει θετικέ απαντήσει στα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε και οι οποίοι θα δουν τι συνθήκε αυτέ από ό,τι φαίνεται να χειροτερεύουν. Η ανάπτυξη δεν γίνεται μόνο, γίνεται μάλλον κυρίω από ισχυρέ επενδύσει, σωστά στοχευμένε επενδύσει που με τη σειρά του δημιουργούν ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ισχυρό και ταυτόχρονα να βρούμε πρόσθετους πόρους ε, για το πλαίσιο αυτό. Δεν θα συζητήσω τώρα τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν για τα ευρωομόλογα και για τον φόρο Τόμπιν. Αλλά για να γίνουν αυτά τα οποία εσεί είπατε κύριε Πρόεδρε χρειάζονται πόροι που δεν υπάρχουν σε αυτή τη φάση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να του βρούμε. Αν πράγματι θέλουμε να κάνουμε τα δίκτυα στον τομέα τη ενέργεια, στον τομέα των μεταφορών, οι διαθέσιμε χρηματοδοτήσει σήμερα είναι χρήσιμε μεν σε ένα κάποιο πλαίσιο και κλίμακα, αλλά δεν είναι επαρκής τουλάχιστον για να ολοκληρωθούν τα προγράμματα αυτά στο σωστό χρονικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε την ιδέα πρόσθετων πόρων επιπλέον του τακτικού προϋπολογισμού. Να πω εδώ ότι δεν τίθεται το πρόβλημα το τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά αντικειμενικά σε έξι μήνες. Ο απολογισμός θα γίνει με βάση αυτά τα οποία θα μπορέσετε να προχωρήσετε αλλά χρειάζεται να υπάρξει γενεοδορία, χρειάζεται να υπάρχει όραμα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ίσως να ολοκληρωθούν σε μια άλλη φάση, αλλά θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει για το κοινό Να Απαιτείται λοιπόν διοργανική συνεργασία, πολιτική συνεργασία και θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό με θάρρος, αλλά και με την ευελιξία που μπορεί να έχει μια μικρή χώρα ενάντια σε μια μεγάλη. Ο κύριος, ευχαριστώ κύριε Κοφέρατη. Ο κύριος Σμιτ θα λάβει τώρα τον λόγο εξ των φιλελευθέρων. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Διατρέχουμε μια δυσχερή περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τρεκλίζει, κλειδονίζεται, εθνικισμός και προστατευτισμός αυξάνονται ως φαινόμενα. Εσείς κύριε Πρόεδρε επομίζεστε σημαντικές ευθύνες και έχετε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσετε όχι μόνο στον οικονομικό τομέα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον χρηματοοικονομικό τομέα, χρηματοπιστωτικό τομέα, στις τράπεζες. Πρέπει να ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση και ε, θα έλεγα δράση. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε την οικονομία της αγοράς. Θα έπρεπε πολύ περισσότερο να ασκούμε επικρίσεις επί των πολιτικών ανδρών που δεν επομίστηκαν τις ευθύνες τους και δεν έδρασαν με υπευθυνότητα. Πολλοί από αυτούς, αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και εδώ παρόντες. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε την πρώτη κατηγορία και την δεύτερη κατηγορία. Την πρώτη ομάδα και τη δεύτερη ομάδα. Εκείνα τα κράτη που ανήκουν στην ε, ζώνη Ευρώπη ευρώ και εκείνα που δεν ανήκουν σε αυτή τη ζώνη. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε λοιπόν το σιδηρούν παραπέτασμα που χώριζε την Ευρώπη σε δύο τμήματα, την δυτική και την ανατολική. Δεν πρέπει να ξαναδιχαστεί ε, ε, η Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο λόγω δύο κατηγοριών κρατών, τη πρώτη και τη δεύτερη, εκείνων που ανήκουν στη ζώνη ευρώ και εκείνων που δεν ανήκουν σε αυτήν. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντα θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι ατυχέστατο το ότι το ίμιση τη Κύπρου δεν εκπροσωπείται εδώ σήμερα. Ελπίζουμε όλοι και θέλουμε Θέλουμε να είναι ενωμένη και ενιαία η Κύπρο και έχετε μεγάλη ευθύνη για να το επιτύχετε αυτό, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για του πράσινου. θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριο Αλφονσί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ω ε, κοσικανός ε, Ευρωβουλευτής, χαιρετίζω την Προεδρία σα που είναι και νησιωτική και μεσογειακή. Λόγω τη κρίση την οποία διανύουμε, πρέπει να ακουστούν οι προσδοκίες αυτού του ζωτικού χώρου για το μέλλον της Ευρώπης, της Μεσογείου. Η κρίση θίγει πολύ την ευρωπαϊκή πλευρά της Ένωσης, την Κύπρο, την Ισπανία, την ε, Νότια Γαλλία, την Ελλάδα. Έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο και έχουμε και ένα κοινό καθήκον να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες ε, των χωρών της γειτονίας μας, όπως εκφράστηκαν τον, την άνοιξη του 2011. Καλύτερη ζωή, ουσιαστική δημοκρατία, και καρποφόρες σχέσεις με την Ευρώπη μέσω των ε, δεσμών που συνδέουν όλους τους λαούς του ευρωπαϊκού χώρου εδώ και αναρρύθμιτα χρόνια. Με πάνω από 90% το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια εκθεσή μου χθε που ζητάει να υπάρξει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη Μεσόγειο. Αυτή η νέα μορφή περιφερική συνεργασία στην Ευρώπη έδειξε όπω και στη Βαλτική ότι είναι δυνατόν οι διάφορε πολιτικέ αναπτυξιακέ τη Ένωση να έχουν ε, καλύτερο αποτέλεσμα συντονισμένε. Πρέπει λοιπόν αυτή η δομή να υπάρξει και στην Μεσόγειο. Έχουμε τώρα ένα νέο προγραμματισμό 2014-2020. Εκεί πρέπει να ενταχθεί για να είναι αποτελεσματική. Πρέπει να δώσουμε στο μεσογειακό χώρο που είναι σε κρίση ένα θετικό μήνυμα. Να υπάρξουν θετικέ πρωτοβουλίε. Και περισσότερη στήριξη χρειάζεται από πλευρά μα. Και θα ήθελα λοιπόν η Κύπρο να, να μπορέσει να αναλάβει τι πρώτε πρωτοβουλίε που θα βοηθήσουν για την περαιτέρω ε, στρατηγική ανάπτυξη τη Μεσογείου. Ευχαριστώ κύριε Αλφονζή. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα στους παρόντες πρόεδρους των ομάδων. Παρακαλώ, όταν ε, γράφετε μόνο ένα λεπτό για τους ομιλητές σας και εκείνοι θέλουν να μιλήσουν, ε, να κάνουν μια ομιλία πέντε λεπτών, είναι αδύνατο για τους διερμηνείς μας να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όταν έχετε ένα λεπτό, να μιλάτε με ρυθμό που να μπορεί να μεταφραστεί. Ευχαριστώ, ο Πασκά, EFD. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ε, ε, η, η Πρόεδρος αναλαμβάνει την ε, Προεδρία σε μια συγκυρία που είναι πολύ περίπλοκη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Κατά το επόμενο εξάμεινο, η Κύπρος δεν θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με τα δικά της προβλήματα, αλλά να συντονίσει και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό θα είναι σίγουρα δυσχερές. Όμως το φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο μας ε, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Χριστόφια καταδεικνύει ότι η Κύπρος έχει προπαρασκευαστεί με πολύ υπεύθυνο τρόπο για την Προεδρία της είναι λοιπόν ε, σε θέση να βοηθήσει να επιτευχθεί πρόοδος στην οικονομική και κοινωνική ζωή στην Ευρώπη. Ένα επιπλέον θετικό είναι ότι η Κύπρος έχει αυτήν την μοναδική γεωγραφική θέση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου. Πιστεύω λοιπόν ότι εφόσον έχετε πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική και επειδή ξέρετε και την κατάσταση στην περιοχή σας, θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε αυτά τα ατού, ούτω ώστε να βοηθήσετε στην επίλυση των πολλών προβλημάτων αυτής της περιοχής. Σας εύχομαι λοιπόν πολύ επιτυχία και σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο ιδιαίτερα υπό το φως συγκεκριμένης ε, ε, γεωγραφικής και ιστορικής σημασίας της Κύπρου. Πρέπει να τονιστεί ότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου τμήμα της επικράτειας βρίσκεται υποκατοχή από τις στρατιωτικές δυνάμεις μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας, της Τουρκίας. Η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει την δημοκρατία της Κύπρου και να επομιστεί τις ευθύνες της μέσα στο πλαίσιο της Τελωνιακής Ένωσης όσον αφορά τα πλοία και τα αεροπλάνα της Κύπρου που θα έπρεπε να μπορούν να, να στα ε, λιμάνια της Κύπρου και στα αεροδρόμια της ε, Κύπρου παρόλο το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Αυτό είναι μια σκανδαλώδης κατάσταση, πραγματικά κατάφορα σκανδαλώδης, όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια που πάντα έλεγε στους πολίτες της ότι οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά την Τουρκία και την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, τροχοπεδούντο αν δεν μπορούσε να έρθει στο ύψο των υποχρεώσεών τη η Τουρκία. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Τούρκο Υπουργό επεσήμανε πρόσφατα ότι δεν συμφωνεί, λέει, για το ότι θα έπρεπε να επιτραπεί, λέει, στην Τουρκία να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα παγώσουν οι ε, διαβουλεύσεις ε, για την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν την ευθύνη να παγώσει τις σχέσεις με την Τουρκία και αυτό δείχνει ότι δεν έχει καμιά αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αξίζει κανένα ε, σεβασμό από τους ε, πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλμπρεχ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της ε, Κύπρου Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Κύπρος και η Πολωνία εντάχθηκαν την ίδια χρονική στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμως ποτέ δεν κάνουμε λόγο για την Κύπρο ως ένα νέο κράτος μέλος αναφερόμαστε υπό την έννοια των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκείνα τα κράτη που βρισκόντουσαν πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα Ποτέ εσείς ε, ως Κύπρος δεν είχατε αντιμετωπιστεί ως νέα χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία λοιπόν να υπάρξει μια γεφυροποίηση, να δημιουργηθεί μια γέφυρα σε σχέση με την Τουρκία και εμάς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία για όλα αυτά τα προβλήματα. Και αναφέρομαι και στις ε, τοποθετήσεις που αφορούν την ε, συνοχή της Ευρώπης με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ω συζητήσει για ένα από τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να βρεθεί η σωστή γλώσσα σε σχέση με την διαμόρφωση των πολιετών δημοσιονομικών πλαισίων. Και ελπίζουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα προ καταλάβει ένα διχασμό, ένα κατακαιρματισμό μεταξύ των κρατών μελών. Ένα διχασμό μεταξύ εκείνων που είναι υπέρμαχοι της συνοχής και άλλων που είναι υπέρμαχοι των δαπανών. Δεν είναι αντίφαση αυτό. Πρέπει να υπερβούμε και να αποφύγουμε αυτή την αντίφαση και να προχωρήσουμε. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε αυθεντικά είναι μεγαλύτερη παραπληρωματικότητα ή συμπληρωματικότητα υπό την έννοια μιας πολιτικής προσέγγισης. Δεν πρέπει να διπλωθούμε διπλασιαστεί το γραφειοκρατικό βάρος και να υπάρξουν επικαλύψεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε χρηστότερη, πιο αποτελεσματική διαμόρφωση των δαπανών. Και γι' αυτό ελπίζω ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι υπέρμαχος και φίλη της ε, καλύτερης διάθεσης των κονδυλίων και της συνοχής. Ευχαριστώ. Κύριε Προεδρεύον, κυρία Κοπά παρακαλώ. Το Συμβουλίου είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η δική σας Προεδρία, αυτό το κρίσιμο εξάμενο του 2012 είναι κομβική κυρίω λόγω των σημαντικών αποφάσεων που η ένωση καλείται να λάβει για να μπορέσει να βγει από την κρίση. θα αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. αρχικά την ίδια την οικονομική κρίση. έχετε τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη να αποδείξουμε στου πολίτε τη ευρώπη ότι θέλουμε και μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να ξαναδώσουμε την ελπίδα σε χιλιάδε νέου που βλέπουν ζωφερό το μέλλον του στου κόλπου τη ένωση. η ανάπτυξη η καταπολέμηση τη ανεργία η δημιουργία θέσεων εργασία είναι τα σημεία στα οποία οφείλουμε όλοι να εστιάσουμε και είμαι σίγουρη ότι εσείς θα το πράξετε με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνη. δεύτερο η σχέση με τη γειτονιά μα. η γεωστρατηγική σα θέση και οι στενέ σα σχέσει με τον αραβικό κόσμο κύριε πρόεδρε σα επιφυλάσσουν ένα σημαντικό ρόλο. η ρευστή κατάσταση στην νότια γειτονιά τη Ευρώπη, οι σφαγέ στη συρία και η ένταση στη μέση ανατολή σα καλούν να αποτελέσετε έναν έντιμο μεσολαβητή ένα διάβλο επικοινωνία και σωστότερη κατανόηση των αναγκών των χωρών αυτών τρίτο το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κανεί σήμερα στην ευρώπη δεν πρέπει να παραλείπει την ανάγκη να ολοκληρωθούν πετυχημένα οι διαπραγματεύσει για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. τέταρτο το ίδιο το σέγγεν. έχετε μπροστά σα την εμπλοκή που δημιουργήθηκε με τη δανική προεδρία στο ζήτημα του σέγγεν και είναι ανάγκη όλων μα να εργαστούμε για να διαφυλάξουμε ένα από τα μεγαλύτερα κεκτημένα και επιτεύγματα τη πορεία μα ο διαμεσολαβητικός σας ρόλος στην ανάγκη να ξεκαθαριστεί πού πάμε θα είναι κεντρικός. τελειώνοντας και πριν ευχηθώ κάθε επιτυχία θέλω να τονίσω κι εγώ με τη σειρά μου την απαράδεκτη στάση μιας υποψήφιας χώρας της τουρκίας απέναντι στην κυπριακή προεδρία με τις δηλώσεις και εγκυκλίους για πάγωμα των σχέσεων της τουρκίας με την προεδρία αυτή η τουρκία οφείλει να δεχτεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και να καταλάβει ότι είτε το θέλει είτε όχι η κυπριακή δημοκρατία δεν μπορεί να παρακαμφθεί αν ειλικρινά επιθυμεί την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. η επιλογή είναι στα χέρια της. ευχαριστώ και εύχομαι πάλι κάθε επιτυχία σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο και σε σχέση με τα, ε, τη δημοσιονομική, τις προσπάθειες από το 2014-2020 για ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ελπίζω πράγματι να στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημα της Κυπριακής Προεδρίας. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν είναι καθόλου εύκολο το εγχείρημα. Μια σειρά ε, χωρών θέλουν περισσότερα κονδύλια. Κάθε χώρα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρία. Χρειάζονται ε, υψηλή, υψηλής αποτελεσματικότητας ικανότητες ε, για να μπορέσει κανείς ε, να δράσει σωστά. Και έχουμε εδώ και συνολικά το 80% ε, του δημοσιονομικού πλαισίου έχει υποβάλει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το σχέδιό της, όμως θα πρέπει να μπορέσουν να υπάρξουν και πιο προθυμένες επενδύσεις όσον αφορά τις υποδομές, τις μεταφορές, όσον αφορά τις επενδύσεις που απαιτούνται και μια σειρά άλλων θεμάτων. Είναι σημαντικό να υπάρξει ανταγωνιστικότητα, να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και να εξαρτώμαστε λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα ε, και δεν πρέπει να γίνει ένα ανατολίτικο παζάρι ε, αυτή η υπόθεση όπου κάθε ένας θα προσπαθεί να αποκομίσει ωφέλης βάρος των άλλων. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, να είμαστε ενωμένοι όλοι μας ε, και στο Ευρωκοινοβούλιο και να μπορέσουμε να εργαστούμε επί των νέων εξουσιών και αρμοδιοτήτων μας ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και να είναι εποφελές το αποτέλεσμα υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ την Κυπριακή Προεδρία για το μήνυμα που μας έστειλε ότι θέλει να εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια κύριο Σαλαβράκος παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε της Ενίας Κύπρου, η μικρή σας χώρα καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της σοβαρότητας των προτεραιοτήτων που προαναφέρετε στην πρωτολογία σας. η ανάπτυξη και η απασχόληση θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ισχυρή ευρώπη. την ίδια στιγμή στη λεκάνη της ανατολικής μεσογείου και στην ευρύτερη μέση ανατολή μια άκρος φωτισμένη περιοχή συντελούνται γεωπολιτικές εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της περιοχής και της ευρωπαϊκής ε, ένωσης οι εξελίξεις στη συρία στο ιράν και η κλιμάκωση των συγκρούσεων αλλά και οι σχέσεις της με την τουρκία μπορεί να πυροδοτήσει ένα ντόμινο εξελίξεων στη μεσόγειο. ταυτόχρονα η κυπριακή προεδρία καλείται να αντιμετωπίσει η προκλητικά υπονομευτική στάση της τουρκίας την οποία καταδικάζω απερίφραστα και καλώ και την ευρωπαϊκή ένωση να το πράξει. αποδοκιμάζω επίσης ότι τμήμα της κύπρου μιας χώρας μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης κατέχεται από ξένο κράτος στρατεύματα της τουρκίας. η κυπριακή δημοκρατία συνηθισμένη στις δυσκολίες έχει τις ευχές όλων μας για να επιτύχει. ευχαριστώ κύριε για την ομάδα του ΕΛΚ ο κύριος Χακμάρκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, οι αξίες της ελευθερίας, της ανοιχτής κοινωνίας και της ελεύθερης αγοράς είναι θα έλεγα τα θεμέλια για την ευημερία αλλά και για τη σταθερότητα την οποία όλοι χρειαζόμεθα και την ανάπτυξη που χρειαζόμεθα. Νομίζω που όπου αυτές οι αξίες αγνοήθηκαν, τα συστήματα είτε απέτυχαν είτε κατεστράφησαν. Αυτό θα πρέπει να είναι λοιπόν το κοινό σημείο εκκίνησης για όλους και για την δική σας Προεδρία. Έχει σημασία να σημειώσει κανείς ότι όπου υπήρξε η αγορά η ελεύθερη της οικονομίας υπήρξε ευημερία και ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια υπάρχει κρίση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυξημένες δαπάνες και ελλείμματα δεν έχουν βοηθήσει την κατάσταση. Αν αυτή θα ήταν η λύση τότε δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Από την άλλη Δεν υποφέρει η Ευρώπη από υπερβολικά ελεύθερες οικονομίες, υποφέρει από υπερβολικά βάρη ρυθμιστικά, γραφειοκρατίες, μονοπόλια και νομίζω ότι ένας από τους πιο βασικούς στόχους και καθήκοντα είναι ακριβώς να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια πλήρως ρυθμισμένη εσωτερική αγορά, ανοιχτή στην επιχειρηματικότητα, ανοιχτή στις επενδύσεις, ανοιχτή στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η πορεία, η πολιτική που θα καταστήσει την Ευρώπη εκ νέου ισχυρή και αυτό θα πρέπει να είναι και ο βασικός στόχος για τη δική σας Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις για την εσωτερική αγορά. Δεν το έχουμε κάνει όσο οφείλαμε, όσον θα οφείλαμε. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι η μεγαλύτερη οικονομία αν θέλετε στον κόσμο αλλά όχι η μεγαλύτερη αγορά. Θα πρέπει εμείς να προχωρήσουμε σταθεροποίηση των οικονομιών, να προχωρήσουμε με την διεύρυνση. Αυτοί όλοι είναι στόχοι που θα δώσουν αποτελέσματα. Περιμένουμε. Κύριε Χακμάκ, η ε, κυρία συνάδελφος Μπερές ήθελε να σας διατυπώσει κάποια ερώτηση. Παρακαλώ κυρία Μπερές. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε, ε, διαβάσατε τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί δεν μιλάμε για οικονομία της αγοράς, μιλάμε για κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι μόνο αυτό που είπατε εσείς για την αγορά και την ελευθερία της αγοράς, αλλά και η κοινωνική διάσταση και ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που αγνοούνται σε αυτή τη φάση. Και όταν μιλάτε για μονοπόλια Έχετε υπόψη σας και τα ιδιωτικά μονοπόλια τα οποία μπορεί να κάνουν τις χώρες να γονατίσουν όπως η Goldman Sachs στην Ελλάδα. Και όταν μιλάτε για την εσωτερική αγορά έχετε μια σφαιρική αντίληψη για την εσωτερική αγορά. Μια πραγματική εσωτερική αγορά που χρειαζόμαστε, που να έχει μια διάσταση εναρμόνισης δημοσιονομική και φορολογική. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Χέκμαρκ, αγαπητοί συνάδελφε. Ε, μου δίνετε τη δυνατότητα να αναπτύξω ακόμα περισσότερο το μήνυμά μου. Καταρχάς, τα μονοπόλια. Η ασδήποτε φύσεως είναι κάτι το αρνητικό που βλάπτει την οικονομία. Και θα συμφωνήσετε, νομίζω, μαζί μου. Όλα τα μονοπόλια, δημόσια μονοπόλια, ιδιωτικά μονοπόλια, είναι καταδικαστέα. Αυτός είναι βασικός θα έλεγα στόχος βασικό χαρακτηριστικό μιας σωστά λειτουργούσης ανοιχτής οικονομίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανοιχτή και να δίνει εναλλακτικέ λύσεις. Δεύτερον, που πρέπει να παρατηρήσω, η οικονομία της αγοράς είναι κοινωνική, γιατί όπου υπάρχουν επενδύσεις, νέες μορφές ανάπτυξης, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και κοινωνική ασφάλιση. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Χάκμαρκα για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο κύριος Φέρμ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και προσβλέπουμε στην Κυπριακή Προεδρία ως επικεφαλής ε, σε σχέση με την σοσιαλδημοκρατική ομάδα ιδιαίτερα σε σχέση με εκείνα τα σχέδια για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, ενδιαφέρομαι όσον αφορά το πλαίσιο για ένα μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για το, τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλο και πιο δυσχερή γίνονται τα πράγματα, διότι κάποιε χώρε επιθυμούν να συρρυκνωθεί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρξουν περικοπές ε, πιστεύουν ότι είναι η μόνη διέξοδος ε, από αυτή την κρίση και οι πλουσιότερες χώρες θα πρέπει από την άλλη πλευρά να υποστηρίζουν ε, τις φτωχότερες χώρες. Κάποιοι όμως φαίνεται ότι δεν φέρθηκαν, δεν ακολούθησαν μια σωστή πολιτική και υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες λέγουν ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί με έναν εθνικό προϋπολογισμό να συγκριθεί όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές, μισθούς κτλ. Όμως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζει την συνιστόσα της αλληλεγγύης. Πρέπει να είναι ένα στρατηγικά αναπόσπαστο κομμάτι της ε, στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ να επιβραδύνετε λίγο, λέει ο πρόεδρο, γιατί δυσχεραίνονται οι διερμηνείς. Λοιπόν, έλεγα ότι σε σχέση με ε, τον στρατηγικό ρόλο που έχουν αυτά τα πράγματα για την Ευρώπη, η προσέγγιση σε σχέση με την ε, ενιαία εσωτερική αγορά που πρέπει να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να ε, μπορέσει να τύχει ολοκλήρωση η Ευρώπη, να υπάρξει καινοτομία και στην έρευνα και στην, και στην καινοτομία. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτή τη στρατηγική και αυτές οι νηστώσεις, Πρόεδρε, για να μπορέσουν να συνενωθούν οι χώρες μας και να οδηγηθούν προς μια ολοκλήρωση, ενώ έχουν τόσες πολλές πολλέ διαφορέ. Πώ μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ενιαία προσέγγιση σε σχέση με τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κ. Ντέιβι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα συγκεκριμένο θέμα θέλω να θίξω. Απευθυνόμενο στον Πρόεδρο. Για να μεταρρυθμίσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική είναι ουσιώδε να υπάρξει μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείριση, ούτως ώστε κάθε ε, αλλιευτικό να έχει σαφείς στόχους για να ανακάμψουν τα αποθέματα. Ορισμένα από αυτά έχουν εκτεθεί από το Κοινοβούλιο, αλλά έχουν παγώσει το Συμβούλιο. Ορισμένα από τα νομοθετήματα προ αυτήν την κατεύθυνση. Το Συμβούλιο δεν τα προωθεί. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαφωνούν όσον αφορά την ε, ερμηνεία τη ε, συνθήκη. Και λογικά επιχειρήματα προβάλλονται και από τι δύο μεριέ. Μπορούν να επιληθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων. Αλλά δεν γίνονται διαπραγματεύσει. Αυτό λοιπόν το αδιέξοδο θέτει εν κινδύνο όλα όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσω τη μεταρρύθμιση τη κοινή ελευτική πολιτική. Ξέρω ότι ο πρόεδρο Μάρτιν Σούλτ το έχει ήδη θίξει. Σα ε, ερωτώ λοιπόν κύριε πρόεδρε, θα αξιοποιήσετε την ευκαιρία να μα πείτε ότι δεσμεύεστε για να αναιρεθεί αυτό το μπλοκάρισμα, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Δεν περιμένω, δεν ζητώ από την Κυπριακή Προεδρία να επιλύσει το πρόβλημα. Σα ζητώ να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει που θα μπορούσαν να επιτύχουν αυτή τη λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Τώρα ο Μάριο Μαύρο. Ευχαριστώ πολύ λέει γερμανικά και συνεχίζει ελληνικά. Ο τύπος της χώρας μου, της Ιταλίας, με ρώτησε θα στηρίξετε την Κύπρο ακόμα και αν ο πρόεδρος είναι κομμουνιστής. Και εγώ απάντησα θα υποστηρίξουμε την Κύπρο Ακριβώς γιατί ο πρόεδρος είναι κομμουνιστής. Κομμουνιστής που εξελέγει δημοκρατικά από το λαό του και η δημοκρατία είναι η βασική θεμελιώδης αξία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερήφανη για τους προέδρους της που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Εσείς κύριε Πρόεδρε ζητήσατε στην ομιλία σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην θέλει να εξάγει συστηματικά το δικό της πρότυπο δημοκρατία. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν θέλουμε να εξάγουμε τη δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να δίδουμε την μαρτυρία της δικής μας δημοκρατίας. Και ο τρόπος με τον οποίο το πετυχαίνουμε αυτό είναι όταν υπενθυμίζουμε στην Τουρκία ότι η στρατιωτική κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου είναι μια μεγάλη αδικία και θα πρέπει οι ίδιοι οι Κύπροι να βρούνε την ιδανική λύση στο πρόβλημά τους. Εμείς δίδουμε τη μαρτυρία μας για την δημοκρατία όταν υπενθυμίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία στις χώρες του νότου της Μεσογείου όπως την Αίγυπτο θα ήταν αδικία να εφαρμόσουν τη Σαρία τον Ισλαμικό νόμο για τα 10 εκατομμύρια χριστιανών κοπτών και να προχωρούν στον ακροτηριασμό των, των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Γι' αυτούς ακριβώς λοιπόν τους λόγους Νομίζω ότι κύριε Χριστόφια θα έχετε μπροστά σας έξι μήνες γεμάτους ενδιαφέρον, γεμάτους αντιθέσεις. Σαν κομμουνιστής που είστε θα θέλετε να ενισχύετε τους εργαζομένους. Αλλά για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να στηρίξετε και τις τράπεζες, οι οποίες σίγουρα τον τελευταίο καιρό έπαιξαν ένα αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη της κρίσης. Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτού του εξαμήνου θα γίνουμε όλοι περισσότερο Κύπροι και εσείς λιγότερο κομμουνιστής. Ευχαριστώ κύριε Μαύρο. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Καταλήν Ιβάν. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς ε, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δεσμευθήκατε να υποστηρίξετε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία την προσπάθειά τους να ενταχθούν στον ε, χώρο Σέγγεν. Ε, διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Χρειαζόμαστε ευρωομόλογα και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να μειωθεί η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, για περισσότερη απασχόληση. Αλλά σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη δημοκρατία περισσότερη προσοχή στο σεβασμό των ε, ευρωπαϊκών αξιών και της δημοκρατίας γενικότερα στην Ευρώπη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια γενικευμένη ιστερία όσον αφορά την δημοκρατία στη Ρουμανία. Ακούσατε τις ε, παρεμβάσεις ε, επ' αυτού σήμερα. Αλλά ήμουν παρόν και όταν μιλήσαμε για τον Περλουσκόνη, για την ελευθερία του τύπου στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, όταν μιλήσαμε για τα λάθη του Ορμπάν και του Μπορισόφ. Οι ίδιοι συνάδελφοι του εκείνη την ε, ε, περίοδο υποστήριζαν τα μέτρα του κυρίου Μπορίσοφ, του κυρίου Ορμπάν, του κυρίου Μπερλουσκόνη. Θα ήθελα να σας πω ότι έχετε καθήκον, αλλά έχετε και τη δυνατότητα να ελέγξετε τι συμβαίνει, ούτω ώστε να υπάρχει σεβασμός στη δημοκρατία στην Ευρώπη και είμαι επισμένο ότι θα ανακαλύψετε ότι η κυβέρνηση Πόντα έχει επιτύχει πολλά για την ελευθερία του τύπου εδώ και δύο εβδομάδε. Ο τύπο δεν είναι απειλή πλέον για την εθνική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κριστίνα Όγιουλαντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Χριστόφια. Καταρχή, θα ήθελα να σα ε, ευχηθώ επιτυχία για να επιτύχετε του στόχου τη ε, Κυπριακή Προεδρία που συμπεριλαμβάνει να ενισχύσετε τι σχέσει με του γείτονε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ελπίζω ότι οι στενέ σχέσει ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρωσία δεν θα γίνουν εμπόδιο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και η επιδείνωση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου πολύ κοντά στη σύνορά μα. Ω εισηγήτρια για την επιβολή κοινών περιορισμών για τι ε, προξενικέ θεωρήσει για του Ρώσου αξιωματούχου που έχουν να κάνουν με την υπόθεση Αργέη Μακνίτσκι, θα ήθελα να καλέσω την Κυπριακή Προεδρία να συμφωνήσει με τη σύστασή μα και να μα βοηθήσει για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και την ασυνδοσία στη Ρωσία. Οι καλέ ε, σχέσει με του γείτονέ μα δεν πρέπει να βασίζονται στην διακριτική και εφεκτική σιωπή. Όταν ε, παρατηρούμε τέτοιε σοβαρέ παραβιάσει του ε, εθνικού και διεθνού δικαίου. Έχετε την ευκαιρία να κάνετε ειλικρινέ και επικοδομητικέ συζητήσει με το Κρεμλίνο και να τονίσετε την ουσιαστική σημασία, την θεμελιώδη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Άντρας Γκιούρκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που ακούσαμε τα τελευταία λεπτά από τους λόγους των προλαλισσάντων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας τα περισσότερα προβλήματα και προσκόμματα τα, θα τα αντιμετωπίσει η Κυπριακή Προεδρία στα δημοσιονομικά θέματα. Η πολιτική συνοχή είναι μεγάλη, τεράστια πρόκληση. Είναι για μας απαράδεκτο τα κονδύλια για την πολιτική συνοχή να περικοπούν, να συρρυκνωθούν. Και αυτό επειδή η πολιτική συνοχή είναι ένα από, ένας τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών πολιτικών και οι όροι υπό τους οποίους διαμορφώθηκαν οι πολιτικές συνοχής ε, εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα σπουδαίοι και σημαντικοί και σε σχέση με όλα αυτά δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η έκφραση της ε, μακροπρόθεσμης αλληλεγγύης ε, και της ενδυνάμωσης αλληλεγγύης. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι επειδή ακριβώς διατρέχει, διανύει μια σοβαρή κρίση η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση η αλληλεγγύη δεν θα είναι μια σημαντική αξία. Θα πρέπει να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες επί των οποίων θα οικοδομήσουμε. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μια μη ισόρροπη κατάσταση. Δεν μπορούμε σε σχέση με τα κονδύλια συνοχή να δεχθούμε περικοπε σε σχέση με την Ουγγαρία, που και μέσω πρόθεσμα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε το 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αν θέλουμε να υπερβούμε με σωστό τρόπο αυτή την κρίση, τότε απαιτούνται τέτοια μέτρα τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω υπερχρέωση, δεν θα οξύνουν την υπερχρέωση. Έτσι θα πρέπει να διαμορφωθεί λοιπόν η πολιτική συνοχή μέσα σε τέτοια πλαίσια. Η Κυπριακή Προεδρία αν μπορεί να υπερασπιστεί, να είναι υπέρμαχος της πολιτικής συνοχής, αυτό θα είναι μείζον και εκτιμένο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Στη συνέχεια ο κύριος Ερτούγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας συγχαίρω που αναλαμβάνετε την ε, Προεδρία και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την εφαρμογή των καθήκων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Πρέπει να εργαστείτε αποτελεσματικά για να υπάρξει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ένωση και ε, αναμένουμε με ενδιαφέρον τις συγκεκριμένες προτάσεις για την καταπολέμηση της ε, ανεργίας των νέων. Το Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει εάν το επιχειρήσετε αυτό. Μεγάλη προτεραιότητα βεβαίως είναι οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και σωστά αναγνωρίσατε και γι' αυτό σας συγχαίρω ότι η χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων θα προσδώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Σας κάνω λοιπόν έκκληση αποφασιστικά να εργαστείτε ούτως ώστε στο Συμβούλιο οι προτάσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Και από αυτό κύριε Πρόεδρε θα μπορούσαν να επωφεληθούν και τα λιμάνια σας ε, στο, στη Λεμεσό και το αεροδρόμιο στην ε, Λάρνακα και η οδός από την ε, ε, Λάρνακα στην Λευκοσία. Φυσικά είναι ανεπίλητο ακόμη, ή μάλλον δεν έχει επιληθεί ακόμη το Κυπριακό. Αλλά κύριε Πρόεδρε, τι σενάριο πρέπει να περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν υπάρξει λύση για το Κυπριακό. Μετά από 38 χρόνια ε, ανεπιτυχών διαπραγματεύσεων γίνεται όλο και πιθανότερο να μην υπάρξει λύση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ. Ως δημοκράτης από την Ολλανδία θέλω να ευχηθώ στον πρόεδρο της Κύπρου κάθε επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο του. Είστε μικρή χώρα. Και εγώ είμαι από μικρή χώρα. Είναι πάντα μεγάλη πρόκληση να κάθεσαι με τους μεγάλους Μέρκελ, Ολάντ, Σούλτς και να προσπαθείς να ε, παίξεις ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ιδιαίτερα με τον κύριο Μπαρόσου που λέει ότι πρέπει να κάνετε προσπάθεια για τα πιο ουσιώδη θέματα. Έχετε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πολλά πρέπει να επιτύχετε σε αυτό. Δεν άκουσα επίσης ε, την λέξη επικουρικότητα σήμερα κατά τις ομιλίες. Πολλά θα πρέπει να κάνουμε εμείς μόνοι μας στις χώρες μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιορίζεται στα κυριότερα θέματα. Φυσικά πρέπει να καταπολεμήσουμε την κρίση, Είπαμε ότι πρέπει να εμβαθύνουμε την ενή αγορά. Αυτά τα αναφέρατε βεβαίως. Αναφέρατε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο βεβαίως. Το αναφέρατε. Αλλά οι εξοικονομήσεις ε, στις οποίες αναφερθήκατε θα έχουν επιπτώσεις ε, στους πολίτες της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη ε, να εξετάσει πολύ προσεκτικά τον προπολογισμό. Όπω είπαν και οι φιλεύθεροι συνάδελφοι, η πολιτική ασύλου Ελπίζετε να ε, επιτύχετε σε αυτήν, να σημειωθεί πρόοδο στο επόμενο εξάμεινο. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα του Σέγγεν και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Υπήρξαν ε, έντονε συγκρούσει για τα θέματα αυτά με το Συμβούλιο και ελπίζω κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα να σεβαστείτε τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επιχειρήσετε να βασιστείτε σε αυτέ για να προχωρήσουμε. Για το θέμα τη Τουρκία, Αναφέρθηκαν πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι περίπλοκο θέμα και είναι πολύ πιο περίπλοκο λόγω των σχέσεων ε, της Κύπρου με την Τουρκία. Με αυτό το υπόβαθρο σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο Σοκράτης, ξέρετε, είπε ότι θα πρέπει όπως και την Αθήνα να αφήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα από ό,τι βρήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για αυτό που είπατε για τον Σοκράτη. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κρίστιαν Βίγκενιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη φιλόδοξη προοπτική που έχετε θέσει και για την ανάγκη που, θα, που υπάρχει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη με τους φτωχότερους πολίτες της. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θα στηρίξουν τις προσπάθειές σας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σας ευχαριστούμε και για τη στήριξή σας για την ένταξη της Ρωμανίας και της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν. Υπάρχει ένας κάποιος συμβολισμός στην Προεδρία σας. Το κέντρο, στο κέντρο της πολιτικής θα είναι μια χώρα η οποία γεωγραφικά βρίσκεται στα απότατα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις μικρότερες ε, ευρωπαϊκές χώρες που θα ηγηθεί της Ευρώπης των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτό δείχνει τη μοναδική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι οι πολίτες μας ίσως κατανοήσουν τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε πετύχει μετά από τις τελευταίες διαβρύνσεις, με την τελευταία διαβρύνση μάλλον. Η γυπνίασή σα, με τον νότο επίσης της Μεσογείου θα υπογραμμίσει την ανάγκη στήριξης των χωρών της περιοχής αυτής στον τομέα της οικονομίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής ανάπτυξης που είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ε, της προσπάθειας να πλησιάσουμε τις χώρες αυτές. Υπάρχει και κάτι άλλο το, το συμβολικό. Μια χώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποδιέρεση θα πρέπει να στηρίξει την ενοποίηση ακόμα και σε επίπεδο δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πετύχουμε επίσης και στα πλαίσια του μελλοντικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και περαιτέρω διευρύνσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Βιγενίνο. Ο κύριος Κούκαν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο Χριστόφια στην Ολομέλεια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσίαση του προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας. Η Κυπριακή Προεδρία αναφέρεται σε κυριότερους άξονες ε, της πολιτικής ώστε να προσεγγίσει περισσότερο η Ευρώπη τους γείτονές της και σε με ιδιαίτερο τρόπο αναφέρομαι στα ανατολικά γειτονικά κράτη και τα κράτη με τα οποία γειτονεύουμε στην περιοχή της ε, Μεσογείου. Και έχει λογική συνέπεια αυτό, διότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου δικαιολογείται αυτή η προσέγγιση και θα πρέπει έτσι να δώσει συνέχεια η Κυπριακή Προεδρία στις προσπάθειες της Δανέζικης Προεδρίας, ε, της Δανικής Προεδρίας όσον αφορά τις προτεραιότητες σε σχέση με την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό πρέπει να τύχει συνέχεια σε σχέση με τις πολιτικές αυτές μελλοντικά. Θα πρέπει να επικεντρωθεί η Κυπριακή Προεδρία στην αναθεώρηση ε, μεταρρύθμιση δράσεων. Ιδιαίτερα έχω υπόψη την καταπολέμηση της διαφθοράς και την καταπολέμηση της ατιμορρησίας Υπάρχουν πολλές χώρες, ε, ε, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, που πλήττονται ιδιαίτερα από αυτές τις μάστιγες. Αν αντιμετωπίζαμε καλύτερα αυτά τα προβλήματα, θα οδηγούσαμε σε μια καλύτερη Ευρώπη. Και αυτό είναι μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στην περιοχή των Βαλκανίων έχει άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια πανευρωπαϊκά, στην ίδια την Ευρώπη. Και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ε, με το Μαυροβούνιο, με την Σερβία, υποψήφιες προς ένταξη χώρες, με τους ηγέτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Όλα αυτά είναι δραστηριότητες μέσα σε ένα πλαίσιο που ε, ε, έτυχε ισχυρών ε, αξιόπιστων θεμελίων και αυτό θα αποτελέσει ένα υφαλτήριο για περαιτέρω δυνατότητες διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσετε προσπάθειες σε όλη αυτή τη συνολική διεργασία. Το να σταματούσαν οι διεργασίες της διεύρυνσης θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των φιλοδοξιών και των στόχων σας. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κούκαν. Και ε, τώρα η κυρία Παπαδοπούλου θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, στη μακραίωνη ιστορία της η Κύπρος γνώρισε πολλούς κατακτητές κι όμως άντεξε σκλαβιές και απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960. Το 2004 με το σπαθί της έγινε μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένεια και το 2008 τη Ευρωζώνης. Σήμερα η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου αν και μικρή σε μέγεθο και διχοτομημένη από του Τούρκου εισβολείς η κύπρος είναι παρούσα και πανέτοιμη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε έτοιμη να αντιμετωπίσει πολλαπλές αντικσότητες την οικονομική κρίση την κρίση χρέους την κρίση αξιών. Είμαστε πεπισμένοι πως η Κύπρος θα τα καταφέρει, γιατί διαθέτει αξιόμαχο ανθρώπινο δυναμικό, γιατί εργάζεται σκληρά και έχει όραμα για μια Ευρώπη των λαών και των αξιών, μια Ευρώπη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αλληλεγγύης. Η Κύπρος είναι πανέτοιμη να προωθήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα, σεμνά, αποφασιστικά και τίμια. Αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη αλληλεγγύη στο νησί μα να αναγνωρίσει το γεωστρατηγικό ρόλο της κύπρου στην ανατολική μεσόγειο. αναμένουμε να ασκήσει περισσότερες πιέσεις στην κατοχική τουρκία να τερματίσει την κατοχή το σφετερισμό περιουσιών τον παράνομο επικισμό και αν δεν το κάνει τότε να τερματίσει την ενταξιακή πορεία της τουρκίας. ελληνοκύπροι και τουρκοκύπροι δικαιούμαστε να ζούμε σε μια ενωμένη πατρίδα. ευχαριστούμε συνάδελφε. Στη συνέχεια η κυρία Θεοχάρους παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκφράζω την περηφάνεια μου για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την πατρίδα μου. Συγχαίρω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια, για την εμπνευσμένη ομιλία του, με την οποία έθεσε ξεκάθαρα τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας από τον πλέον επίβολο, αυτό του, του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι τον πλέον ανθρώπινο της επισητιστικής βοήθειας για αυτούς που πεινάνε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Βάτσον, μπορεί η Κύπρος να είναι μοιρασμένη, αλλά δεν είναι μισή όπως μας λέει ο κύριος Μπαΐς και αν είναι μοιρασμένοι τα σειρματοπλέγματα στο νησί μα τα έφερε η απεικιοκρατική δύναμη η βρετανία η οποία δυστυχώ παραμένει στον τόπο μα με την αναχρονιστική μορφή των βρετανικών στρατιωτικών ε, βάσεων. και για τα δεινά που υφίστανται οι ελληνοκύπροι και οι τουρκοκύπροι σήμερα το μέγιστο μερίδιο τη ευθύνη φέρει ο τουρκικό κατοχικό στρατό, ο οποίο στη συνέχεια τη απεικιοκρατία κρατά το νησί μοιρασμένο Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο Σούλτς γιατί έθεσε αποφασιστικά σταθερά και δίκαια την υπόθεση της προκλητικής τουρκικής στάσης των Ήβρεων και της ε, προσβολής προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Το έθεσε επιτακτικά στην Άγκυρα. Έθεσε την Τουρκία πρώτων ευθυνών της όχι μόνο για τη στάση της έναντι της Κυπριακής προεδρίας αλλά και έναντι της τάσης της κύπρου συνολικά έναντι της κυπριακής δημοκρατίας διαχρονικά. γι' αυτό νομίζω και θέτω και εγώ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενώπιον των ευθυνών του οφείλουμε και εμείς να πάρουμε μια απόφαση για άμεση διακοπή των ενταξιακών συνομιλιών της τουρκίας εάν η χώρα αυτή δεν συμμορφωθεί. ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα έχει το λόγο ο κύριος ε, Αλεχάνδρο Κέρχας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Χριστόφια, σας εύχομαι κάθε επιτυχία, μεγάλη επιτυχία στην Προεδρία σας και στις φιλοδοξίες σας για να εργαστείτε για μια Ευρώπη περισσότερο ολοκληρωμένη και δίκαια. Συμμερίζομαι τις απόψεις που εσείς εκφράσατε στην δική σας εισαγωγική παρατήρηση, διότι πραγματικά χρειαζόμαστε μια πιο υγιή οικονομία, για μια κοινωνία που θα είναι πιο υγιής. Δεν θα υπάρξουν οικονομίες υγιής με άρρωστες κοινωνίες, άρρωστες λόγω αδικίας, λόγω έλλειψης κοινωνικής ολοκλήρωσης και μη έκφρασης αλληλεγγύης. Ως προς όλα αυτά βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία στην Ήπειρό μας είσαστε πρόεδρος μιας μικρής χώρας, μπορεί να είσαστε όμως ε, ε, πρόεδρος μιας επιτυχούς μεγάλης προεδρίας και αυτό σας εύχομαι για την ολοκλήρωση, για την δυνατότητα κυκλοφορίας των εργαζομένων, για την οδηγία απόσπασης ε, εργαζομένων, για το corporate aid, για τους εποχιακά εργαζόμενους. Υπάρχουν μυριάδες εργαζόμενοι στην Ευρώπη που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους και απομονωμένοι λόγω της, και μέσα σε μια παγκοσμιοποίηση. τα φυλάκια. θα ήθελα να δραστηριοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε με κάθε ενεργητικότητα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Στη συνέχεια Κέλαμ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για μένα η Κύπρος είναι η πεμπτουσία ενός πολιτισμικού και ιστορικού θαύματος. Ασσύριοι, Πέρσοι, Πέρσες, ε, Ρωμαίοι, ε, άλλοι κατέκτησαν την ε, νήσο. Όμως επιβίωσαν οι Κύπροι και διασφάλισαν και διατήρησαν την ταυτότητά τους μέσα σε ένα πλαίσιο ζωντάνιας και δημιουργικότητας. Ξεκινώντας αυτή την ιστορική σημασία προεδρία σας, είναι καλό να θυμόμαστε τα λόγια του Προέδρου Μπαρόζο. Μπορούμε να επιτύχουμε αν είμαστε ενωμένοι όλοι μας. Όχι αν ένας των άλλων. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους στόχους μας από κοινού. Ένας από τους πρώτους στόχους της ε, Κυπριακής Προεδρίας θα πρέπει να είναι η ανάκτηση και ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης ε, των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκλείστηκε από την λήψη αποφάσεων όσον αφορά το Σέγγεν. Την προηγούμενη εβδομάδα μονομερός το Συμβούλιο άλλαξε σημαντικές πτυχές ε, και άρθρα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Πώς μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι λοιπόν για την ανάγκη περισσότερης Ευρώπης όταν το ένα θεσμικό όργανο ε, δημιουργεί μη σώροπες σχέσεις μεταξύ ε, άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στόχος για την ολοκλήρωση λοιπόν της ενιαίας εσωτερικής αγοράς δέκα ετών διάρκειας. Θα πρέπει εδώ να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τα προσκόμματα τα οποία οποία Ζητώ από την Κυπριακή Προεδρία όχι μόνο να δώσει συνέχεια με την εμβάθυνση των προσπαθειών για την ενιαία εσωτερική αγορά, αλλά να υποβάλει και ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο πρόγραμμα για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την ενιαία εσωτερική αγορά ε, με την άρση των εμποδίων και προσκομμάτων. Θα πρέπει επίση να προαχθεί η ψηφιακή ενιαία εσωτερική αγορά και να χρησιμοποιηθεί ω κλειδί για να απελευθερωθεί το δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπέρ τη δημιουργικότητα και της ανάπτυξης. Και τέλος θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι είναι μια ανώμαλη κατάσταση να έχουμε συνομιλίες και διαβουλεύσεις με μια υποένταξη χώρα που ε, έχει υποκατοχή ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνες μας για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πρόεδρο, σας ευχαριστώ συνάδελφε. Η συνάδελφος Φλασικόβα Μπένοβα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ευχηθώ μια σωστή Προεδρία, μια ευχάριστη Προεδρία και να πω ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς Βλέπω ότι ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματός σας προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση της κρίσης και θα ήθελα να μάθω πώς η χώρα σας ε, αντιμετωπίζει τα δύο μέσα καταπολέμησης της κρίσης, δηλαδή το θέμα της καταπολέμησης των ε, φορολογικών παραδείσων και το θέμα της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης. Ξέρω ότι εσείς περιμένετε βοήθεια από το Ταμείο Σταθεροποίησης και οι υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν με τη βοήθεια αυτή. Και εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι κάτω του 800 ευρώ. Οπότε θα πρέπει να εξηγήσω στους εκλογείς μου πώς μπορούμε να στηρίξουμε μια χώρα σαν τη δική σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο Ράιμερ Μπέργκε στη συνέχεια παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε Χριστόφια, εύχομαι στην Κυπριακή Προεδρία σας κάθε επιτυχία στο έργο της προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της Κύπρου. Συχνά μικρότερες χώρες ε, είναι καλύτεροι και πιο έντιμοι διαμεσολαβητές από τι μεγαλύτερες χώρες ε, και τείνουν να λάβουν υπόψη και τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περισσότερο και με τις πρώτες συζητήσεις με τον ε, κύριο Υπουργό Μακογιάννη και για τα θέματα των πολιτών δημοσιονομικών πλαισίων πολλά μπορούμε να δούμε ότι υπόσχονται αυτές ε, οι προσπάθειες και σε σχέση με τις συζητήσεις και για όσον τη Δευτέρα για τη στενότερη συνεργασία και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκπόνηση αυτών των πολιτών δημοσιονομικών πλαισίων με αυστηρή τήρηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπω απορρέουν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτά τα χαιρετίζουμε και με ιδιαίτερο τρόπο τα καλαδεχόμαστε. Και θα ήθελα να προσθέσω ευχαρίστω εδώ ότι για μα αυτή τη συζήτηση η έκθεση της ειδική Επιτροπής εξακολουθεί να αποτελεί τα ενδεδειγμένα θεμέλια. Χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των κονδυλίων προ όφελο τη στρατηγική του 2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια αυθεντική στρατηγική και δράση ώστε να μπορέσουν επιτέλου οι στόχοι τη συνθήκη Λισαβόνα να επιτευχθούν. Είμαστε υπέρ της, του ενιαίου χαρακτήρα του προπολογισμού και είμαστε πρόθυμοι να προβούμε σε, σε βάθο συζητήσει που θα αξίζουν αυτό το, το όνομα, το χαρακτηρισμό προτού καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο συμφωνία για τα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια. Διότι θέλουμε να συμφωνήσουμε για το αποτέλεσμα και όχι να μα σερβίρουν ένα αποτέλεσμα χωρί να έχουμε εμπλακεί και για το οποίο θα μπορούσαμε μόνο καταψηφίσουμε κατά τα τέλη του έτου. Σα εύχομαι καρποφόρα και γόνιμη συνεργασία υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπέγκε. Στη συνέχεια κυρία Εστρέλα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Χριστόφια, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Την χρειαζόμαστε αυτήν και για την ανθεώρηση της ε, οδηγίας ε, για την γονεϊκή ε, άδεια, μητρική άδεια που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το, το 2010 ως εισηγήτρια και μέχρι σήμερα το Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε στα δικά μας αιτήματα και προτάσεις ούτε εξέφρασε ενδιαφέρον στο να υπάρξει ένας διάλογος έστω και άτυπος για να εξευρεθεί μια ισόρροπη λύση που θα εξυπηρετεί τις ευρωπαϊκές οικογένειες. Η κρίση ήταν ένα πρόσχημα και για την αντιμετώπιση της ε, μητρικής άδεια ε, ως, ένας, ε, ως ένα ελάσσονο σημασίας, ίσονος σημασίας θέμα. Υπάρχουν χρήματα και κονδύλια για τις τράπεζες αλλά όχι για τους πολίτες. Περνάμε μια πολύ σημαντική κρίση και αυτή είναι η δημογραφική κρίση. Όλο και πιο υπερήλικος γίνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, πράγμα το οποίο διακυβεύει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και την ίδια την οικονομική ανάπτυξη. Αναμένουμε και προσβλέπουμε στο ότι η Κυπριακή Προεδρία θα μπορέσει να αποτροχ αυτό το θέμα, να το απελευθερώσει και να μπορέσουν να ληφθούν τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπόψη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Συνάδελφε, στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κ. Γκαρίγα Πολέδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένας από τους ε, συναδέλφους μας στην ε, δική σας πολιτική ομάδα ο οποίος δυστυχώς έχει χάσει τη ζωή του, ο Μιγγέλ Πόρτας και εγώ ήμασταν συγητές για τα θέματα αυτά. Δεν συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, συμφωνήσαμε όμως στο γεγονός ότι τα διαρθωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι η λοκομοτίβα της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ε, τα 55 λοιπόν αυτά δισεκατομμύρια ευρώ των διαρθρωτικών ταμείων που είναι ανα προγραμματοποιήσιμα έχουν ενσωματωθεί στο λεγόμενο σχέδιο ανάπτυξης. Αλλά δεν υπάρχουν δυνατότητες για διαφορετικά ταμεία ή για ανάπτυξη αν δεν υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις πληρωμών. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει αρκετά ποσά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον αναπρογραμματισμό των διαφορετικών ταμείων. Και αυτό γιατί τον Νοέμβριο του 2011 η συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου απέτυχε. <clears throat> Δεν κατέληξε σε συμπέρασμα. Για τον προϋπολογισμό του 2013 τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει μια αύξηση 6,8% για τον προϋπολογισμό και εσείς προτείνετε μόνο 2,9%. Πιστεύουμε λοιπόν ότι Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, εμείς θέλουμε να μπορέσετε να συμβιβάσετε αυτά τα δύο τόσο δύσκολα και διαφορετικά στοιχεία όπως είναι η πίεση της Κομισιόν για περισσότερα χρήματα και η αντίδραση των κρατών μελών που δεν θέλουν περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να δεχτείτε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ρούιμπικ. να ευχαριστήσω τον κύριο Γκαρίγκα γιατί ακριβώς το θέμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει για μας αποφασιστικής σημασίας. Κύριε Γκαρίγκα, θεωρείτε ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει σε κάποια τμήματα αυξηθεί από τα κράτη-μέλη και μειωθεί σε κάποια άλλη ότι είναι επαρκής αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκαρίγκα Ποϊέδο. κύριε Ρούμπικ. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, όπως και εγώ φυσικά, ποιε είναι οι θέσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 και πόσο αποκλίνουν από τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε όπως και εγώ ο ίδιος ότι χωρίς επαρκείς πόρους για πιστώσει πληρωμών δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δεσμεύσει που έχει αναλάβει το Συμβούλιο για το σχέδιο, για το Σύμφωνο Ανάπτυξης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει να διαδραματίσει ένα αποφασιστικό ρόλο, όχι μονάχα όπως είπε ο κ. Μπέργκε για τις δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά και για να απεμπλέξει τον προϋπολογισμό του 2013. Αν παραμείνει στο αδιέξοδο προϋπολογισμός του 2013 δεν μπορεί να υπάρχει Σύμφωνο ανάπτυξη και Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό έχει κομβικό ρόλο η Κυπριακή Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω 10 αιτήσει για να λάβουν το λόγο. Οι βουλευτές δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω σε όλους το λόγο γιατί έχουμε και ένα άλλο σημείο στην ημερησία διάταξη το οποίο ακολουθεί πριν από τη διαδικασία ψηφοφοριών. Ζητώ την κατανόησή σας λοιπόν. Ο κύριος Κουμουτσάκος είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα κύριε πρόεδρε της κυπριακής δημοκρατίας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η ανάληψη της προεδρίας του ευρωπαϊκού συμβουλίου είναι ιστορικά πολιτικά και συμβολικά κορυφαία στιγμή για την κυπριακή δημοκρατία. η ούτως ή άλλως απαιτητική άσκηση καθηκόντων της προεδρίας αυτό το εξάμεινο σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής και ευρύτερης κρίσης γίνεται μια πραγματική πρόκληση. η ευρώπη οφείλει ενωμένη και αλληλέγγυα να βρει το βηματισμό της να ξαναβρει την ψυχή της να αποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ευρωπαίους πολίτες. στην επίτευξη αυτού του υψηλού στόχου καλείται να συμβάλει αποφασιστικά η κυπριακή προεδρία απερίσπαστη από τις γνωστές απαράδεκτες προκλήσεις αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής θεσμικής τάξης και των ευρωπαϊκών θεμελιωδών αρχών από μια υποψήφια χώρα. κύριε πρόεδρε μην παρασυρθείτε. αφήστε αυτή την χώρα στην ευρωπαϊκή μοναξιά που έχει η ίδια επιλέξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε κύριος Χαιρετίζω την ανάλυση της Προεδρίας από την Κύπρο παρά το ότι βεβαίω θα είναι δύσκολο το έργο σας με το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Βεβαίω υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η χρήση των μέσων συνοχής τα οποία περιορίζονται. Υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα την πατρίδα μου, την Ουγγαρία η οποία κινδυνεύει από το ότι 20-30% των κονδυλίων της συνοχής χάνονται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από το πλαφόν να ορίσουν και ένα κατώτατο όριο και αυτό μπορεί να το κάνει η Κυπριακή Προεδρία. Το έχει κάνει η Δανέζικη Προεδρία και ήθελα να παρακαλέσω την ε, Κυπριακή Προεδρία να ολοκληρώσει αυτό το οποίο μέλησε να κάνει η Προεδρία της Δανίας ε, μια ανακοίνωση να πει δηλαδή πως είναι απαράδεκτο να χάνει η Ουγγαρία 20-30% των κονδυλίων της συνοχής. Σας ευχαριστώ. Βάγγελ είναι τώρα στον καταλογό μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την σοφία την οποία μοιραστήκατε μαζί μας λέγοντας πως δεν θα πρέπει να εξάγουμε τις δικές μας ιδέες και αντίληψη για την κρίση. Βεβαίως αναμένουμε πολλά από την Κύπρο όταν μιλάμε για τομείς κρίσιμους όπως ε, η Μέση Ανατολή, αλλά γνωρίζουμε πως η Κύπρος είναι διάσημη για τη διπλωματία της. Επίσης ε, Ε, ο κύριος ε, Κασουλίδης ήταν ε, επικεφαλής αυτής για κάποιο καιρό και είχε αντιδράσει μάλιστα θυμάμαι σε μια ομιλία του κυρίου Γκρέχαμ Βότσον. Πρέπει να πω πως δεν επικροτούμε την τουρκική στάση ως προς την Κυπριακή Προεδρία. Η Τουρκία νομίζω θα μπορούσε να είναι πιο λογική αν ήμασταν κι εμείς κάπως πιο ανοιχτοί. Και εσείς που είστε μια μικρή χώρα μπορείτε να κάνετε πολλά για την ευρωπαϊκή προοπτική άλλων χωρών όπως και η Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος κρατάει ζωντανή την ε, παράδοση του Αποστόλου Παύλου και Βαραβά. Έχουμε μια κτηνόδη τουρκική κατοχή ενός ε, μέρους της ε, νήσου. Αλλά βεβαίως η Κύπρος ε, κοιτάει και προς την κατεύθυνση της Μόσχας. Και εσείς κύριε Πρόεδρε δάσατε στην Μόσχα και ξέρετε βεβαίως πως έχει τις γνωστές διαθέσεις ο Πούτιν. Κύπρος για οικονομική στήριξη θα πρέπει να στραφεί στην Ευρώπη. Τα σημαντικά ζητήματα είναι η επίβλεψη που ασκεί η Κύπρος στις τράπεζες στην χώρα της. Πώς μπορεί οι τράπεζες αυτές να έμπλεξαν τόσο πολύ. Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τους στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Τέλος, να σας ε, ευχηθώ καλή δύναμη και τις ευχές μου για την Προεδρία σας. Ο κύριος Ρώση, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κύπρος ε, είναι ε, ένα καθίστο πλευρό της Ευρώπης. Ε, δεν επέβαλε στην Τουρκία η Ευρώπη να απελευθερώσει τη Βόρεια Κύπρου που δέχτηκε την εισβολή το 1974, αλλά τη χρηματοδοτεί. Ο κυπριακό πληθυσμό του Βορρά είδε να του παίρνουν τα σπίτια, τη δουλειά, τη θρησκευτική ελευθερία. Λοιπόν, είχατε και απαγορεύτηκε να πάει, να πάει στα κατεχόμενα για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Ε, και έχουν καταστραφεί διάφορα μνημεία ε, θρησκευτικά. Ε, θα ήθελα το εξάμεινο τη Κυπριακή Προεδρία να μπορέσει να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διηγηθεί σε αποφάσει κατά των εισβολέων και τελικά να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών του και όχι των μικρών ισχυρών ε, οικονομικά που θέλουν να έχουν σχέση με τη Βόρεια Κύπρο. Σα εύχομαι κύριε Πρόεδρε να κάνετε κάτι για τη γη σα και για, τους, για το λαό σας που αξίζει να μπορεί να επιστρέψει να είναι ε, ιδιοκτήτης στα σπίτια του. Κυρίω στα σπίτια του. Herr Ευχαριστώ κύριε Μιλώντα για ανάπτυξη και απασχόληση, το μιλάμε μόνο, δεν μπορούμε να τα εξασφαλίσουμε. Μεγαλύτερη αιτία για την ανεργία στην Νότια Ευρώπη είναι ε, το ευρώ. Ε, και, αυτοί που, και θα πρέπει να σωθούν αυτοί που θέλουν να μείνουν εκεί. Τελικά η παγκοσμιοποίηση και συμφωνίε, με αναδυόμενε συμφωνίε έχουν καταστρέφουν ε, την βιομηχανική μα βάση και πετάνε του Ευρωπαίου εργαζομένου από τι θέσει του. Η νέα Προεδρία αναφέρεται στη δημογραφική αλλαγή υπό τη μορφή του γυράσκοντο πληθυσμού και αναφέρεται στις αναγκαίε απαντήσει για την καταπολέμηση του φαινομένου. Ποιες μπορεί να είναι άραγε αυτές οι απαντήσει, Χρειάζεται να βλέπει κανείς το μέλλον να έχει καλή μεταναστευτική πολιτική και καλύτερη ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών που προέρχονται από διάφορους πολιτισμούς ε, και εθνοτικό ιστορικό. Οι νέοι του τρίτου κόσμου θα αντικαθιστούν τους ε, Ευρωπαίους που δεν γεννώνται. Ε, κανονικά αυτό θα γινόταν. Αλλά τι θα κάνουν αυτοί που θα έρθουν, θα φέρουν τον τρίτο κόσμο μαζί τους και θα μεταμορφώσουν τμήματα της Ευρώπης στον τρίτο κόσμο. Οι διακεκριμένοι λαοί δεν είναι προϊόν διακεκριμένων πολιτισμών. Οι διακεκριμένοι πολιτισμοί, οι διαφορετικοί πολιτισμοί είναι προϊόν διαφορετικών λαών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η Κύπρος έχει το πιδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις. Μια από αυτές είναι να, το, να περατωθούν οι διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι να καταλήξουμε σε ουσιαστικούς προϋπολογισμούς που να ευνοήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση ιδίως των νέων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όμως πρέπει να έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση Ιδίω στις πολιτικές οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξη και της, αποτελεσμα... και απασχόλησης και την πολιτική συνοχής δηλαδή και την πολιτική καινοτομία. Εγώ έρχομαι από μία από τις θαλάσσιες περιοχές της ε, Πολωνίας και είμαι σίγουρος ότι θέλετε να δώσετε μια νέα όθηση στην θαλάσσια πολιτική της πολωνιας και ειμαι σίγουρο οτι Ένωσης. οθηση στην θαλασσια πολιτικη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. καθε επιτυχια σα εύχομαι. Ευχαριστώ κύριε. κύριος Σας ευχαριστώ. Καλύτερη Ευρώπη είναι το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας που είναι το όνειρο όλων των πολιτών της Ευρώπης. Ανησυχούν όμως οι πολίτες για την οικονομική κρίση και το χειρότερο κομμάτι της κρίσης ελπίζουμε να το έχουμε περάσει. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Φοβάμαι πως όπως και οι προηγούμενες προεδρίες οι περισσότερες προτεραιότητες ε, θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ε, πίσω από την οικονομική κρίση. Θέλουμε να πιστέψουμε τις διαβεβαιώσεις Προεδρίας πως ε, τα προβλήματα των Κυπριακών Τραπεζών δεν θα επηρεάσουν την Κυπριακή Προεδρία. Όμως μπορεί να προκληθούν προβλήματα για την συνένεση στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω πως δικαίως συμπεριέλαβαν τις εθνικές προτεραιότητες οι κυπριακές αρχές, δηλαδή τη θαλάσσια πολιτική, και την ασφάλεια στη θάλασσα. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως γιατί έχουμε στο, στην, στο πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 χώρες με κοινή μοίρα και αν ε, το πλοίο ανατραπεί θα πνιγούμε όλοι. Καλή επιτυχία λοιπόν εύχομαι. Γκέι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπαρόζο όμως είπε χτες πως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 2,9 δι ή 4,9% του ΑΕΠ. Αλλά είχαμε 40,4 ε, δισεκατομμύρια που δόθηκαν σε στοιχεία ενεργητικού και πάνω από 100 δισεκατομμύρια συνολικά από το 2008. Οπότε εδώ πέρα δεν μπορεί να λέει ο Γάιδαρος στον πετνό κεφάλα. Όλοι στην ίδια μοίρα είμαστε. Ευρωζώνη, Ηνωμένο Βασίλειο, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βοηθήσουμε ε, λοιπόν ο ένας τον άλλον και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Και ελπίζω η Κυπριακή Προεδρία γιατί μέχρι τώρα, από τώρα μέχρι το τέλος της δεν θα έχει την Προεδρία κάποια μεγάλη χώρα, θα συνεργαστεί για να καταπολεμήσει την τάση την διακυβερνητική και πρέπει να θυμόμαστε πως τον προηγούμενο αιώνα 60 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σκοτώθηκαν στους πολέμους. Έχει πέσει το τείχος του Βερολίνου. Εάν λοιπόν ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση μπορούμε να πούμε πως είχαμε μια χρυσή εποχή στην Ευρώπη. Παρατάτε λοιπόν τη μάχη κατά της διακυβερνητικής προσέγγισης. Σας ευχαριστώ κύριε Μίτσελ, έχετε μία μπλε κάρτα. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ, θα συμφωνείτε μαζί μου πως είναι πολύ σημαντικό να δίνει σαφεί δηλώσει κομισιών. Για τα σχόλια λοιπόν του κυρίου Μπαρόζο χτε για τα 64 δις λίρες βρετανικών κονδυλίων που πλήρωσε η τότε σοσιαλιστική κυβέρνηση στις τράπεζες. Να σας πενθυμίσω πως 30 δις από αυτά, τα μισά σχεδόν, πήγαν για να διασώσουν Ιρλανδικές και Ολλανδικές τράπεζες, βρετανικά λεφτά. Και σκοπεύει το Ηνωμένο, σκόπευε το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκρίνει τις ε, προτινόμενες συμφωνίες για τη μεταρρύθμιση των τραπεζών, αλλά κατόπιν προτάσεων της Γαλλίας και άλλων κατέβηκε η φιλοδοξία αυτών των προτάσεων. Γιατί επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο ήθελε επίσης να διαχωρίσει λιανικές και επενδυτικές τράπεζες και αυτό σχεδόν αδύνατο το έχει καταστήσει η ε, Κομισιόν. Συμφωνείτε λοιπόν ως προς αυτά και τις ε, προτεραιότητες υπερχόμενες προεδρίας. Απάντηση. Πράγματι αναγκαίο είναι και θα θυμάστε βεβαίω πως η μικρή ε, Ιρλανδία δέχεται περισσότερες εισαγωγέ από το Ηνωμένο Βασίλειο από όσο ε, εξάγει στην Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία μαζικά, το οποίο μας δείχνει πώς χρειάζεται ένα τον άλλον και όπως είπα δεν πρέπει να λέει ο γάδαρος στον πεντινό κεφάλα. Κλείνω τώρα τη διαδικασία Catch the Eye και ερχόμαστε τώρα στι καταληκτικέ παρεμβάσει τη Κομισιόν και του Συμβουλίου και καλό καταρχήν τον Επίτροπο κύριο Σεφκοβιτ να λάβει το λόγο. σα. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε Χριστόφια, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συζήτηση αυτή κατέδειξε σαφώς ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσατε κύριε Πρόεδρε για την Κυπριακή Προεδρία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και καλόδεκτο. Επίσης είναι γεγονός ότι η Προεδρία σας έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στον οικονομικό και, και πολιτικό στίβο. Είναι σαφέ από αυτή τη συζήτηση ότι η πρώτη προτεραιότητα θα είναι η για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο τα μέτρα ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κρίσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης και η καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς. Ας πω λοιπόν δύο λόγια για τις κέρυες αυτές προτεραιότητες, ιδίως για τις πολιετή δημοσιονομικές προοπτικές, Ακόμα και μετά από αυτή τη συζήτηση, είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε σε όλου ότι δεν πρόκειται για ένα προπολογισμό για τι Βρυξέλλε ή για το Στρασβούργο. Είναι ένα προπολογισμό ο οποίος δείχνει ποια είναι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία για τους πολίτες της Ευρώπης, για τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητε στην Ευρώπη. Η σωστή λοιπόν αντιμετώπιση των δαπανών θα πρέπει να λάβει υπόψη το ότι 94% των δαπανωμένων ποσών επανερχόνται στις χώρες, στις περιφέρειες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια προσθέμενη αξία η οποία δεν μπορεί πάντα να προκύψει σε εθνικό επίπεδο προϋπολογισμού. Είναι λοιπόν μία από τις καλύτερες επενδύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει την ευφυα ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Όταν μιλάμε όμως για ευφυα ανάπτυξη δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό χωρίς τον προϋπολογισμό που εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ιδίως την υποστήριξη σχεδίων και προγραμμάτων σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης. Μιλάμε τώρα για μια Ευρώπη των 27 και σύντομα των 28, μια προσέγγιση χρειάζεται να διατηρήσει και την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να τη θυσιάσουμε στο βωμό της οικονομίας γιατί αυτή η συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική ιδίω για τα κράτη-μέλη τα οποία δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι η κρίση κατέληξε σαφώς ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και βαθύτερη οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση και χρειαζόμαστε να έχουμε και ένα οδικό χάρτη προς την ε, πολιτική ένωση ξεκίνησε η διαδικασία αυτή από το Συμβούλιο με την Τραπεζική Ένωση γιατί είναι ο πιο πιεστικός στόχος και αυτός ο οποίο είναι εφικτό σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς αλλαγή των συνδικών. Και εξάλλου είναι απαραίτητη μια τέτοια κίνηση για να επαναφερθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τους νέους τραπεζικούς κανονισμούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολύ περισσότερα από άλλα μέλη των G20. Για την ενιαία αγορά παραμένουν πολλά βέβαια τα οποία πρέπει να πράξουμε. Η άρση των εμποδίων θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ μας. Πρέπει να δράσουμε λοιπόν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Έχουμε λοιπόν κάθε ελπίδα ότι η Κυπριακή Προεδρία θα μπορέσει να επιτύχει συμφωνίε στα θέματα αυτά μέχρι το τέλο του χρόνου για συμφωνίε που έχουν να κάνουν με δημόσιε προμήθειε, με επαγγελματικά προσόντα και άλλα μέτρα τα οποία θα τονώσουν την ανάπτυξη και τα οποία έχουν εντοπιστεί στι αρμόδιε εκθέσει εφέτο. Θέλω να υπογραμμίσω και πάλι την ε, ανάγκη μιας συνεκτικής αντιμετώπισης για τα πολιετή δημοσιονομικά θέματα για την νομοθετική διαδικασία και για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό με την κοινοτική, με την ενωσιακή μέθοδο και ελπίζω ότι θα παραμείνει αυτό και ο κύριος άξονας της Προεδρίας σας. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε λοιπόν από τα μέλη του Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταδείξουμε καλύτερα ότι θέλουμε να πετύχουμε και μπορούμε από κοινού να πετύχουμε, κύριε Πρόεδρε. Πολλοί ομιλητέ έχουν ήδη εκφράσει την ικανοποίησή τους για την πλήρη προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας και την δήλωση της απόλυτης αποφασιστικότητό σα να επιτύχετε στο εγχείρημα αυτό. Η Κομισιόν θα σταθεί στο πλευρό σα να σα βοηθήσει, γιατί <clears throat> αυτό θα είναι και ο καλύτερο στόχο για του Ευρωπαίου πολίτε. Θέλω λοιπόν να σα ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία σα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Αντιπρόεδρο για την παρέμβασή του. Δίνω τώρα το λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Χριστόφια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φίλες και φίλοι, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω θερμά τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων για τα καλά τους λόγια για την Κυπριακή Προεδρία και την προετοιμασία της χώρας μας για να ασκήσουμε τον ρόλο του Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Αυτό είναι για μας πολύ σημαντικό και είναι ενθαρρυντικό αντιλαμβάνεστε. Είναι ενθαρρυντικό γιατί εκπροσωπούμε μια μικρή χώρα η οποία φιλοδοξεί να υπηρετήσει ανιδιοτελώς την Ένωση χωρίς καμιά εθνική σκοπιμότητα χωρίς να θέλει να προωθήσει δικά της συμφέροντα. Για τον απλό λόγο ότι είναι μια μικρή χώρα, είναι νέο μέλος της Ένωσης και όπως είπαν και διάφοροι ομιλητές, οι Κύπροι έχουν φιλότιμο και είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τιμήσουν και την χώρα και την Ένωση. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Διαπιστώνω φυσιολογικά και μια γκρίνια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η γκρίνια προέρχεται από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πρώτα απ' όλα τα οικονομικά, τα κοινωνικά, ως Ένωση και ως ξεχωριστές χώρες. Πώς είναι δυνατόν να την αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ενωμένοι. Θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ στενά τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και αυτά που είπα στην εισαγωγική μου ομιλία δεν είναι σχήματα λόγου χωρίς τη συνεννόηση και την καθημερινή επαφή μεταξύ των θεσμικών οργάνων δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτε μα τίποτε απολύτως. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε, να ρίχνουμε ευθύνε κάποιοι στο Συμβούλιο, κάποιοι στην Επιτροπή, κάποιοι θα λένε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τα λέει καλά και αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ένωση των συμβιβασμών. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Διότι εκπροσωπούμε διαφορετικές χώρες, ενίοτε και διαφορετικά συμφέροντα. Εμείς, ως ένας έντιμος και αντικειμενικός διαμεσολαβητής, θα προσπαθήσουμε να μπούμε στη μέση για να συμβιβάσουμε θέσεις, απόψεις και πολιτικές αν θέλετε. Εμείς επιχειρούμε κάτι καινούριο. Να παντρέψουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι κάτι, θέλω να πιστεύω, καινούριο. Ας το δοκιμάσουμε, γιατί τα μέσα που δοκιμάσαμε μέχρι σήμερα μας παίρνουν και πιο βαθιά στην κρίση. Και αυτό δεν είναι προς τιμή της Ένωσης. Οι λαοί περιμένουν πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κυπριακό λαός, όταν αποφασίσαμε όλοι ομόφωνα ότι θα εντάξουμε τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επανηγύρισε και ανέπνευσε έτσι ελεύθερα θα έλεγα γιατί θα μπαίναμε σε αυτήν την μεγάλη οικογένεια και έβλεπε έναν καλύτερο μέλλον. Ε, αυτή τη στιγμή όλοι οι λαοί, οι απλοί άνθρωποι δεν βλέπουν μπροστά τους αυτόν το καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να προβληματιστούμε. Εμείς δεν εισηγούμαστε κομμουνιστικές πολιτικές και θέλω αυτό να το σχολιάσω ιδιαίτερα διότι αναφέρθηκαν ο κομμουνιστής πρόεδρος κλπ. Ναι, είμαι αυτός που είμαι και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που είμαι. Και γιατί προέρχομαι από έναν κόμμα το οποίο υπηρετεί 90 χρόνια τον Κυπριακό λαό, υπηρετεί τη δημοκρατία, ενώ σε θύματα υπερασπιζόμενων της δημοκρατίας, μαζικά πήρε μέρος στον πόλεμο κατά του φασισμού, θύματα πολλά, υπερασπίστηκε τη δημοκρατία στη διάρκεια του πραξικοπήματος, αγωνίστηκε με ειρηνικά μέσα για απαλλαγή από την απεικιοκρατία, ε, πρόσφερε στους εργαζόμενους καλύτερες συνθήκες ζωής. Είναι μπροστάρι σε αυτό το κόμμα μου. Γι' αυτό ανεξαρτήτως τι έγινε στη Σοβιετική Ένωση ή στις οποιασδήποτε άλλες χώρες, εγώ μπορώ να μιλώ για το ΑΚΕΛ, μπορώ να μιλώ για την Κύπρο και για τον εαυτό μου ως ένα αγωνιστή για τη δημοκρατία. Τα πέντε χρόνια τα οποία κυβερνούμε τη χώρα νομίζω είναι, είναι αποδεικτικό στοιχείο αυτών των γεγονότων. Ένιωσε ο κύριος Κασουλίδης ή ο κύριος Μαυρονικόλας ή η κυρία Θεοχάρους ποτέ να μειώνονται ή να καταπατούνται τα δημοκρατικά δικαιώματα του κυπριακού λαού στην διάρκεια αυτής της προεδρίας. Ένιωσαν οι φίλοι τα 7 χρόνια που προέδρευε ο Χριστόφιας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ήταν απέναντι στα έδρανα οποιαδήποτε καταπάτηση των δικαιωμάτων τους αντίθετα. Αντίθετα λειτουργεί απόλυτα η δημοκρατία στην Κύπρο και είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Κατά συνέπεια μην ανησυχείτε ότι ο κομμουνιστής θα κάνει ζημιά στην Ένωση. Ο κομμουνιστής θα προσπαθήσει για μια καλύτερη Ένωση με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό το λέω και θα το παλέψω στα πλαίσια πάντοτε των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα κάνουμε επανάσταση, μη φοβάστε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά στην Κύπρο για τον Κυπριακό, θέλω να πω στον κύριο Βότσον, με τον οποίο συζητούμε εδώ και χρόνια για τον Κυπριακό, γιατί είναι μέλος και της ομάδας επαφής με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ότι δεν πρέπει να απευθύνεται σε μένα και να με καλεί να συνομιλήσω με την Τουρκία. Πρέπει να απευθυνθείτε στην Τουρκία κύριε και να τους πείτε συνομιλήστε με τον Χριστόφια. Διότι αρνούνται να συνομιλήσουν με τον Χριστόφια. Και εδώ είναι έτσι υποκατηγορία η Τουρκία για λόγους αρχής αν θέλετε. Λέω στον κύριο Ερτογάν, κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ δεχτείτε με να συνομιλήσουμε διότι έχω ένα όραμα το οποίο θέλω να σας αναλύσω που αφορά και τους Ελληνοκύπρους και τους Τουρκοκύπρους και στο κάτω-κάτω συμφέρει και στην Τουρκία η υλοποίηση αυτού του οράματος. Εγώ δεν τρέφω τα οποιαδήποτε εχθρικά αισθήματα απέναντι στον τουρκικό λαό. Αντίθετα, είμαι συναγωνιστή με τους Τούρκους α, απλούς ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και σήμερα στην Τουρκία των αλλαγών και του εξυγχρονισμού διότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τούρκων, των Κούρδων και των διαφόρων άλλων κοινοτήτων στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, θέλω να το τονίσω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την άποψή μου για λόγου αρχή, σύσσωμη, θα έπρεπε να καταδικάζει κάθε ενέργεια τη Τουρκία, η οποία υποβαθμίζει το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ενός κράτους, όχι απλώς μέλους της Ένωσης, μέλος, μέλους όλων των διεθνών οργανισμών, με πρώτον και καλύτερα τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι πανέτοιμος. Τα πέντε χρόνια της Προεδρίας μου είναι χρόνια συνεχούς, ανελειπούς, ακούραστης προσπάθειας να υπάρξει διάλογο και λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω, όταν αναλάμβανα να δώσω τη μάχη για να εκλεγώ πρόεδρο και είχα αντίπαλο μου το φίλο μου το Γιαννάκη, λοιπόν, έκανα μια ξεκάθαρη δήλωση. Και η δήλωση μου ήταν ότι ο πρώτος, αν όχι ο αποκλειστικός λόγος που διεκδικώ την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να εργαστώ σκληρά έχοντας υπόψη τις καλές μου σχέσεις με πολλούς τουρκοκύπριους και πολιτικά κόμματα τουρκοκυπριακά να εργαστώ λοιπόν σκληρά και ακούραστα για επανένωση της πατρίδας μας. Γιατί εγώ είμαι υπέρ σίγουρα της ειρηνικής συμβίωσης και της αδελφικής συνεργασίας των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Η Κύπρος ανήκει στους Κυπρίους Είτε αυτοί είναι Ελληνοκύπροι, είτε είναι Τουρκοκύπροι, είτε είναι Μαρονίτες, είτε είναι Αρμένιδες, είτε είναι Λατίνοι. Βλέπετε είμαστε μια πολυπολιτισμική χώρα, εν πάση περιπτώσει, και επειδή είμαι λίγο διεθνιστής, τι να κάνουμε, οι κομμουνιστές είναι και διεθνιστές. Λοιπόν, ε, θέλω όλοι μαζί να εργαστούμε για το καλό του τόπου μας, ως αφέντες της πατρίδας μας. Ούτε οι Βρετανοί έχουν θέση στην Κύπρο, ούτε οι Τούρκοι έχουν θέση στην Κύπρο, Ούτε οι αδελφοί μας οι Έλληνες με την κακή έννοια έχουν θέση στην Κύπρο. Θα πρέπει να αφαιθούμε ελεύθεροι και να είστε σίγουροι ότι τότε θα έχουμε σχέσεις προνομιακές και με την Τουρκία και με την Βρετανία και ασφαλώς και με την Ελλάδα. Προνομιακές θα είναι οι σχέσεις. Και πολύ στενές και πολύ καλές θα είναι αυτές οι σχέσεις. Αυτή είναι η δική μου υπόσχεση προς τον Κυπριακό λαό την οποία επαναβεβαιώνω και ενώπιον αυτού του ωραίου σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό μου. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από την Τουρκία. Γιατί υπάρχουν επεκτατικές πολιτικές από πλευρά της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο και επεκτατικές βλέψεις. Και λυπούμε που το δηλώνω αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της Συρίας μου. Ξέρω ότι μετά το τέλος τη Συρίας δεν θα επαναδιεκδικήσω την προεδρία της δημοκρατίας μέχρι το τέλος της θητείας μου στην τελευταία στιγμή να αγωνίζομαι ακούραστα για την επανένωση της πατρίδας μου. Και βεβαίως και για μια ένωση η οποία να είναι ένωση για τους πολίτες της, για τους λαούς της Ευρώπης. Έχουμε μια καυτή πατάτα στο χέρι μας. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις, αλλά εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Ένα είναι η ελευθερία της αγοράς και άλλο είναι η ασυδοσία της αγοράς. Εγώ είμαι ενάντια στην ασυδοσία της αγοράς και θέλω να σας το δηλώσω με παρησία. Χρειάζεται παρέμβαση και από τις κυβερνήσεις οι οποίες εκλέγονται από το λόγο για να κυβερνήσουν. Δεν μπορεί να μας κυβερνούν οι αγορέ. Πρέπει να κυβερνήσουν οι κυβερνήσει που δημοκρατικά εκλέγονται από τον λαό. Λοιπόν, υπόσχεση ότι όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί έχουν καταγραφεί, δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα ασφαλώ, έχουν καταγραφεί, υπάρχουν σημαντικότατες εισηγήσει και προτάσει, τι οποίε δεν μπορεί παρά να λάβουμε σοβαρά υπόψη και σε συνεργασία με τον πρόεδρο Σούλτ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον πρόεδρο Μπαρόζο, θα προσπαθήσουμε να βρεθούν οι λύσεις εκείνες οι οποίες θα υπηρετήσουν καλύτερα την, τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμότατα που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ θερμότατα, επαναλαμβάνω, για τις θέσεις και τις παρατηρήσεις τις οποίες έχετε θέσει, τις οποίες θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε για τις ευθύνες ε, που αναλαμβάνετε. Καλή επιτυχία και ελπίζουμε να έχουμε και καλή συνεργασία.